speak Czech or is it? No, English is not so good. so good. Czech is possible. Yeah, all Yeah. Okay, uh, no problem for you. No, no, Czech but, okay. but Best for you. Dobré odpoledne. Vítám všechny kolegy. Καλώς ορίσατε, λέει ο Πρόεδρος. Καλώς όρισαν όλοι οι συνάδελφοι εδώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής βιομηχανίας, ενέργειας. Και θα πρέπει να σας πω ότι η κυρία ε, Σατορή απουσιάζει η πρόεδρος. Όπω ξέρετε, πάντοτε το αεροδρόμιο των Βρυξελών επιφυλάσσει κάποιε εκπλήξει. Οπότε, εάν δεν έχετε αντίρρηση, θα την αντικαταστήσω εγώ. Και τώρα, κύριε Σωτήραξη, τη σημερινή μα συνεδρίαση. Επίση, θα πρέπει να καλωσορίσω τον Υπουργό, τον κύριο Γιάροσλαβ Νεβέρβιτς, Λιθωνός Υπουργός Ενεργείας. Μας τιμά με την επίσκεψή του. Οπότε, και ακούτε, ακούτε την ε, μετάφραση από τους Δερμηνείς. Λειτουργεί η Δερμηνία. Ναι, ναι, α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επομένως, γιατί δεν έχετε αντίρρηση, χωρίς να πούμε τίποτα άλλο προκαταρκτικό, θα τους ευθύς αμέσως τη σκητάλη εις τον Λιθουανό Υπουργό για να προβεί εις μία εισήγηση ενός ε, τετάρτου. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε τι έχει να μας πει ή στα πλαίσια της ε, κυκλική Προεδρίας που είχε αναλάβει. εδώ και σας ευχόμαστε καλή δύναμη, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία υπό αυτή σας την ε, ιδιότητα, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι αναλάβατε την ε, Προεδρία επί ένα εξάμεινο, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολα θέματα με των οποία να εργαστούμε έχουμε ε, τον ε, προϋπολογισμό για το μέλλον και ε, μου είναι το, το έργο της Επιτροπής μας και επομένως έχετε τη σκετάλη Καλώς ορίσατε και πάλι κύριε Υπουργέ. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, είναι για μένα μεγάλη τιμή που μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω το πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας ενώπιον σας, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Λιθουανία είναι η πρώτη χώρα της Βαλτικής που θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Υπουργών το επόμενο διάστημα. Αυτό αποτελεί μεγάλο προνόμιο αλλά και μεγάλη ευθύνη. Χαίρομαι που τώρα αφού παρουσιάσαμε το πρόγραμμα της Προεδρίας, θα, αφού παρουσιάσω το πρόγραμμα της Προεδρίας, θα έχω τη δυνατότητα να συζητήσω ε, μαζί σας θέματα σημαντικά και για την Επιτροπή σας αλλά και για όλους τους ε, πολίτες της Ευρώπης. Όλοι γνωρίζουμε, λέει ο, ο Υπουργός στα Αγγλικά, ότι το Κοινοβούλιο βρίσκεται στο επίκεντρο της ε, δημοκρατικής διαδικασίας της Ευρώπης και ότι η στενή συνεργασία της Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα με, για στην Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας τα θέματα ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Λιθουανική Προεδρία ως εκ τούτου θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για μια επιτυχημένη συνεργασία ώστε να παραμείνει ανοιχτή και, δια... να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει επίσης προτεραιότητα στα αποτελέσματα. Ελπίζω ότι, μπορεί... μπορούμε μαζί να οικοδομήσουμε πάνω στην εξαιρετική δουλειά που επετεύχθη κατά τη διάρκεια της ε, ελληνική, της Ιρλανδικής Προεδρίας για να πετύχουμε περισσότερους στόχους του προγράμματος αυτού της Προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μακρόπνοες αποφάσεις τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και σήμερα αντιμετωπίζουμε ακόμα την, την επίγουσα πρόκληση της δημιουργίας ανάπτυξης και θέσεων εργασίας κυρίως για τους νέους. Οι προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας αντικατοπτρίζουν αυτές τις δυσκολίες όπως και το όραμα μιας ανοιχτής και ε, παγκοσμίως υπεύθυνης Ευρώπης. Αυτές οι προτεραιότητες θα είναι και οι τρεις πυλώνες της Προεδρίας μας, δηλαδή αξιόπιστη, αναπτυσσόμενη και ανοιχτή Ευρώπη. Αξιόπιστη σημαίνει ότι θα μπορέσει να προσφέρει οικονομική σταθερότητα και καλά δημόσια οικονομικά, υγιή δημόσια οικονομικά. Χρειαζόμαστε την ανάπτυξη που θα οδηγήσει πραγματικά θέσεις εργασία. Θα ήθελα να παρουσιάσω εν τα βασικά ενεργειακά ζητήματα που θα τεθούν επιτάπητο στη Λιθουανική Προεδρία. Η ολοκλήρωση τη εσωτερική ενεργειακή αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2014 είναι βασική μα προτεραιότητα. Έχουμε δεσμευτεί σε αυτό το στόχο και επειδή θα έχει οικονομική και ε, προσφορά όπως επίσης και η επίπτωση της ασφάλειας του εφοδιασμού θα επηρεάσει την ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς. Ο στόχος είναι επίσης σημαντικός για τα θέματα που αφορούν τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη της Ένωσης για την επίτευξη της κλιματικής αλλαγής και των ενεργειακών στόχων του 2020. Είναι ευπρόσδεκτη έκθεση για την ε, εσωτερική αγορά σε ενέργεια του κυρίου Μπούσεκ, η οποία συζητήθηκε από την Επιτροπή σας και θα, ε, και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ε, επίσης η δουλειά μας θα στηριχθεί σε αυτό και στην ανακοίνωση της Επιτροπής κάνοντας ε, την, εσωτερική αγορά ενέργειας να λειτουργήσει όπως επίσης και το πρόγραμμα δράσης καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 7 Ιουνίου. Αυτά τα συμπεράσματα αυτά τα συμπεράσματα αντιμετωπίζουν το ρόλο και τα δικαιώματα των καταναλωτών, των ευάλωτων καταναλωτών, το θέμα των, των ρυθμιζόμενων τιμών. Το Δεκέμβριο η Προεδρία θα, αναφερθεί, θα αναφέρει στην ε, κατάσταση στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας η ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης ε, της ενεργειακής πολιτικής είναι ο δεύτερος πυλώνας της προτεραιότητας της Λιθουανικής Προεδρίας στον ενεργειακό τομέα. Καθώς ε, είναι όλο και πιο αλληλένδετες η εσωτερική και η εξωτερική αγορά, χρειαζόμαστε σταθερή και ε, διαφανή ενεργειακή αγορά για να εξασφαλίσουμε ασφάλεια στον τομέα της ενέργειας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά την προμήθεια ε, από εξωτερικές, εξωτερικούς προμηθευτές. Μόνο με συνεργασία και με αλληλεγγύη μπορούμε να δώσουμε στην Ένωση τη δυνατότητα να μιλάει με μια φωνή απέναντι σε εξωτερικού εταίρου, την ενίσχυση τη διαπραγματευτική μα θέση. Μια έκθεση για την υλοποίηση τη ε, ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια ε, εφοδιασμού ενέργεια και για την διεθνή συνεργασία προβλέπεται στα, από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2011 και κυρίως αναφέρεται για τον ε, Συμβούλιο Συμβούλιο του Μαΐου 2013. Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω την, ε, την ε, ε, πολύτιμη δουλειά του κυρί, της έκθεσης του κυρίου Χερτσόγκ σε σχετικά με την συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής με εταίρους πέρα από τα σύνορά μας. Ε, δεδομένων των μεγάλων σημαντικών εξελίξεων που έχουν το μεταξύ συμβεί στον τομέα των εξωτερικών ενεργειακών σχέσεων, η Λιθουανική Προεδρία με τη βοήθεια της Επιτροπής θα αναθεωρήσει και θα ενημερώσει τις κατευθύνσεις που τέθηκαν από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2011. Αυτό θα ενισχυθεί από το Ενεργειακό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τώρα όσον αφορά το σχέδιο οδηγίας για την έμεση αλλαγή χρήση γης, είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόοδο που έγινε στη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα αποτελέσει ισχυρή βάση για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι έντονες διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο στη διάρκεια του προηγουμένου εξαμήνου έχουν ενισχύσει την άποψη ότι η έμεση αλλαγή χρήσης γης από την προαρρογή βιοκαυσίμων είναι σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ε, η, ε, η έκθεση πρόοδος της Κομισιόν για την ε, ανώσιμη ενέργεια που ε, δημοσιεύτηκε φέτος τον Απρίλιο δείχνει ότι τα κρατημέλη προχωρούν καλά στην επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων αλλά επίσης δείχνει ότι η δυσκολία συνεχίζεται καθώς η πορεία γίνεται δυσκολότερη προς το τέλος τα Συμβούλια Ενέργειας και Περιβάλλοντος τον Ιούνιο ε, έλαβαν υπόψη τους τις συζητήσεις και τις ε, εναλλακτικές της, σε σχέση με την έμεση αλλαγή χρήσης γης και ε, έχουν μας αφήσει να αποφασίσουμε για τις κατευθύνσεις της, κατευθύνσεις μελλοντικής δουλειάς. ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις κοινέ συζητήσεις μας. Η εντύπωσή μου είναι ότι τα τρία θεσμικά όργανα εκτιμούν κατά τον ίδιο τρόπο την ανάγκη να περιοριστεί η έμεση αλλαγή χρήση υγιής από τη μία, ενώ ταυτόχρονα θα, θα διατηρούνται οι σαφείς προ, ε, επενδυτικές προοπτικές και θα μπορέσει να, επιτευχθούν, να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπό την έννοια αυτή θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή σας. Ε, με βάση όλα αυτά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε το θέμα. Το πλαίσιο του 2030 για τις πολιτικές του κλίματος και της ενέργειας αφορά την ανάπτυξη στρατηγικής που ξεπερνά τους στόχους του 2020. Στηρίζεται στους δικούς χάρτες του 2050 και θεωρεί τον καλύτερο τρόπο για τη χρήση της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί, αποκτήσουμε οικονομία ανταγωνιστική, βιώσιμη και ασφάλεια όπως επίσης και ένα ενεργειακό σύστημα ε, ε, το να βλέπει τα πράγματα μακροπρόθεσμα είναι χαρακτηριστικό στον τομέα της ενέργειας ε, λόγω του, του μεγάλου χρόνου ζωής της υποδομής ή και λόγω του ότι αυτό έχει, ε, κάθε πράξη συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα λόγω της υποδομής της. Ταυτόχρονα οι επενδυτές χρειάζονται προβλεψιμότητα στο θεσμικό πλαίσιο. πρέπει να γνωρίζουμε πού θα βρισκόμαστε μέχρι το 2030 τον τρόπο και καθώς θα έχει, ε, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί εδώ και μόνο μια εβδομάδα η διαδικασία διαβουλεύσεων που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές πλευρές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο ενέργειας και κλίματος στο μέλλον. Οι στόχοι. Ε, θα, θα πρέπει να είναι δεσμευτική η στόχοι κλίματος και ενέργειας για το 2030 και αν ναι ε, θα πρέπει να είναι και για τις ανανεώσιμες ενέργειες και για την εξοικονόμηση ενέργειας λόγω των νομικά δεσμευτικών μέσων που υπάρχουν και πρέπει να γίνει αναθεώρηση πριν από το 2020. τα μέσα πολιτικής. Ποια είναι τα κατάλληλα μέσα ε, η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια εφοδιασμού είναι σημαντικά θέματα και ε, δεν μπορεί να αναπτύσσεται σε απομόνωση η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιθουανική Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης. Είναι σαφές κυρίως ότι θα πρέπει να, ε, να επιστρέψει η ανάπτυξη και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις απαιτήσει της ανταγωνιστικότητας. Πώς θα πάρουμε υπόψη μας τις δεσμεύσεις των εταίρων μας σχετικά τον περιορισμό της επιπτώσης στο κλίμα. Ε, πώς μπορούμε επίσης να εξασφαλίσουμε καλή, σωστή διανομή των προσπαθειών ε, που θα εξασφαλί, ανάμεσα στα κράτη-μέλη και πώς θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο τις ε, διαφορετικές επενδυτικές δυνατότητες των βιομηχανικών κλάδων και των ομάδων καταναλωτών. Θα ήθελα τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού. Η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει τη μια δημόσια διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο και τώρα ε, προετοιμάζει τις αξιολογήσεις τις ε, μελέτη επιπτώσεων για κάθε κράτος μέλος. Η Λουθανική Προεδρία θα διερευνήσει τη δυνατότητα οργάνωσης της παρουσίας αυτών των αποτελεσμάτων. Το θέμα αυτό θα είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του επόμενου μήνες και απαιτείται συνήθεια συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε επίσης ότι το σχέδιο κανονισμού για την και η γνωστοποίηση των επενδυτικών έργων στον τομέα των υποδομών ενέργειας μπορεί να ολοκληρωθεί στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Αυτό απαιτεί αλλαγή της νομικής βάσης και ζητώ με τη συνεργασία σας και συγκεκριμένα την, βοήθεια της εισηγήτριας κυρίας ε, Βαλεάν. Το Συμβούλιο υπογρήμασε στα συμπεράσματά του για, τις ανανεώσιμες για την ανανεώσιμη ενέργεια τον περασμένο Δεκέμβριο ότι η αναμενόμενη αύξηση στη χρήση βιομάζας για σκοπούς που αφορούν την ενέργεια τα επόμενα χρόνια ενισχύει την ανάγκη να θεωρηθεί η βιώσιμότητα των διαστάσεων αυτών από τη χρήση της βιομάζας η, Ευρω... η... τελευταία έκθεση για την βιωσιμότητα της βιομάζας από πλευράς Κομισιόν παρουσίασε σύμφωνα με την ε, Οδηγία για τις Ανανόσιμες Ενέργειες τον αριθμό, των έναν αριθμό συστάσεων προς τα κράτη-μέλη που έλαβαν υπόψη στην ανάγκη να αποφευθεί η εμφάνιση πιθανώς ε, ασυμβίβαστον μεταξύ τους προγραμμάτων. Περιμένουμε την ε, πρόταση που υποσχέθηκε η Κομισιόν για τις απαιτήσει της βιωσιμότητας για την ε, στερεή και αέρια βιομάζα, τον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψήξη. Ε, ενώ έχουμε να μελετήσουμε την πρόταση πριν την σχολιάσουμε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων των ανανεώσιμων και όχι να προσθέσει αβεβαιότητα στο ε, ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο Ενέργειας θα πρέπει να μελετήσει την απόφαση το Δεκέμβριο. Η ανακοίνωση για την ενεργειακή τεχνολογία και καινοτομία συζητήθηκε στο Συμβούλιο Ενέργειας του Ιουνίου σε μια συζήτηση πολιτικής όπου συμφωνήθηκαν οι κατευθύνσεις που στηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν. Ε, εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποβάλει την ανάλυση της για τα στοιχεία και τους παράγοντες που κατευθύνουν τις ε, τιμές ενέργειας και το κόστος όπως έχει ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαΐου για την ανταγωνιστικότητα. Η Λιθωνική Προεδρία θα είναι έτοιμη να διευκολύνει μια συζήτηση επί της πολιτικής στο ε, ε, Συμβούλιο Ενέργειας του Δεκεμβρίου. Όσον αφορά τα θέματα πυρηνικής ενέργειας, θέλω να αναφερθώ στην αναθεώρηση της οδηγίας του 2009 για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, που θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στον τομέα αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διευκολύνουμε τις επικοδομητικές συζητήσεις με το Συμβούλιο. Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας είναι ζωτική σημασία για όλους τους Ευρωπαίους. Αναγνωρίζουμε πλήρως τη σημασία της επίτευξης στόχων που θα αφορούν τις, τις συνθήκες λειτουργίας των υπουργενικών εγκαταστάσεων. Η προκαταρτική δουλειά θα ξεκινήσει στο Συμβούλιο σε ένα σχέδιο πρότασης που έχει υποβάλει η Κομισιόν εδώ και ένα μήνα και το οποίο είναι ευπρόσδεκτο. Επίσης προσβλέπω στη, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να σας επισημάνω τα βασικά ε, ε, ε, τις βασικές εκδηλώσεις της Προεδρίας με το υπόλοιπο του έτους. Άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Βίλνιους 19 και 20 Σεπτεμβρίου μια υψηλού επίπεδου διάσκεψη για θέματα ενεργειακής υποδομής που θα δώσει έμφαση στην εφαρμογή του καταλόγου PCI της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, οικοδόμηση ενός ε, ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου 4-5 Νοεμβρίου και επίσης θέλουμε να σας υποδεχτούμε στο Βίλνιους στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής σας 15-17 Ιουλίου. Και τέλος δεν ζητάμε συγνώμη για, για τα δύσκολα θέματα που έχουμε θέσει στη Λιθουανική Προεδρία. Αυτό περιμένουν από εμά οι πολίτες μας. πιστεύουν πιστεύω ότι θα πρέπει και θα κατα... Ε, να καταφέρουμε και πράγματι θα καταφέρουμε πολλά αν συνεργαστούμε στενά και ε, αποτελεσματικά. Η εμπειρία και η γνώση τη Επιτροπής σας είναι, είναι πολύτιμη στον τομέα, στην προσπάθεια αυτή. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μαζί σας και με τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο καθώς ε, όλοι μας προσπαθούμε να πετύχουμε του κοινού στόχου στον τομέα τη ενέργεια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Děkuji vám, pane ministře, za velmi εμείς ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την εισήγησή σας. Ήταν πάρα πολύ ενδελεχής και μας εξηγήσατε το πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Η Επιτροπή μας συζητά και έχει αρμοδιότητα για θέματα ενεργείας. Θεωρούμε ότι αυτό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σπουδαίο ως πολιτική. Και πάλι σας την επαγγελματική, παρουσίαση και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. τυχόν να σας θέσουν. Θα πρέπει να μιλήσει για τρία λεπτά. Έχω το λόγο οι συνάδελφοι τώρα. Πρώτα πρώτα η κυρία Γιόρνταν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Εμείς στην ιστορική αγορά έχω μια ερώτηση σε σχέση με την ιστορική αγορά. Ξέρουμε ότι ε, έρχεται το 2014, οπότε έχουμε πάρα πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Πολλέ προκλήσεις πριν φτάσουμε το 2014. Πώς λογαριάζει η Προεδρία να πείσει τα κράτη-μέλη ε, να εφαρμόσουν το τρίτο ενεργειακό πακέτο μέτρων μέχρι το τέλος ενός έτους. Είπατε ότι θα το πράξετε αυτό, αλλά ακριβώ τι θα κάνετε. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω όσον αφορά τις ε, υποδομές σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική. Θα χρειαστούμε δέκα λέγαμε στην αρχή. Όμως ε, τώρα ξέρουμε ότι για να συνειδητρώσουμε τα χρήματα που χρειάζονται πρέπει να ελκύσουμε επενδυτέ. Το θέμα είναι πώς θα τους ε, ελκύσουμε, πώς θα τους πείσουμε να επενδύσουν τα χρήματα που έχουμε ανάγκη. Τι λέτε, Τώρα, σε αυτή την οδηγία για την ποινική ασφάλεια, μας μιλήσατε για το έργο το οποίο έχετε επιτελέσει στο Συμβούλιο, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, συζητούμε την ίδια οδηγία. Είναι θέμα συναπόφαση, οπότε γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί η θετική εργαστή συνεργασία. Οπότε για πέστε μας πώς θα προχωρήσετε, πώς θα εξασφαλίσετε την ανοιγία συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Τελευταία σημαντικό, θα πρέπει να μιλήσουμε για την ε, ενεργειακή πολιτική με ορίζοντα του 2030. Εσείς πώς βλέπετε αυτόν τον ορίζοντα. Είστε ικανοποιημένο με το πλαίσιο που έχει γραφτεί για το 2020 και απλώς θα το παρατείναμε το 2030 ακριβώ το ίδιο ως έχει ή θα πρέπει κάτι να μεταβληθεί. Ο Πρόεδρος. Ας υποβληθούν έξι ερωτήσεις και κατόπιν έχουμε τις απαντήσεις. Μην απαντάτε μία-μία τις ερωτήσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ. Ε, είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Και επίσης ε, εκτιμώ ιδιαίτερα και αυτό που είπατε, έστω και κάπως ε, γενικά, ε, σχετικά με τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα για τη βιομάζα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πραγματί κάποια διευκρινήση σχετικά με τους χρήστες της ε, βιομάζας. Θα πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση και στην πρώτη θέση θα πρέπει να έχουμε την ε, επεξεργασία των ε, ζωοτροφών. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει βέβαια και η ε, βιο, βιομηχανία, όπως τα έλεγα, και αυτή θίγεται σε δεύτερη φάση, διότι ακριβώς αυτή η βιομηχανία είναι εκείνη η οποία εκμεταλλεύεται την μοριακή δομή της βιομάζας και κατόπιν τούτη η βιομάζα για αυτήν είναι πολύ σημαντική. Το τρίτο που ενδιαφέρει είναι η ενέργεια. Όσον αφορά τη βιομάζα, μπορεί να σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος και αναφέρομαι κυρίως στην ε, άμεση μετατροπή της επιρόλησης ε, την βιομάζα σε αέριο και επίσης ε, στη δυνατότητα το αέριο αυτό να το εκμεταλλευόμαστε. Άρα δηλαδή υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες ε, είναι εν λειτουργία και πιστεύω ότι πάνω σε αυτή τη βάση πράγματι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ενεργειακά τη βιομάζα χωρίς καύση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε τις βασικές πηγές ε, ρήπανσης της ε, ατμόσφαιρας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσο μπορείτε να δεσμευτείτε σχετικά με όλα αυτά γιατί αν μπορούσαμε να τα επιτύχουμε αυτά θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα ευρώς ε, για τη χρήση της βιομάζας, ε, για την παραγωγή ενέργειας αλλά και, και για την διαφύλαξη της καθαρότητας της ατμόσφαιρας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χάλ. Πάρα πολύ θετικό θεωρώ το ότι αναφέρθηκε ο στόχος του ορίζοντα 2030 και τώρα που πρέπει να τα εν ώψη αυτού του ορίζοντα και να δούμε τώρα κατά πώς το καταφέρει πριν από το τέλος του έτους ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωση, με λευκή βίβλο κάτι το οποίο θα έρθει στην ώρα για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 12 Δεκεμβρίου. Δεν θα ενθαρρύνετε εσείς να γίνει μια συζήτηση για το πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Αυτό το οποίο είναι μια προϋπόθεση για να γίνει η συζήτηση για τον οριζόντα του 2030. Σε σχέση με την αυτάρκεια της προμήθειας, ε, την ύπαρξη αποθεμάτων κλπ. Όπως το να πετύχει η Επιτροπή. Άρα, θα πρέπει να δεν κατι μέλη σε σχέση με το τι μπορούν να πετύχουν και όχι αναγκαστικά με τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τώρα όσον αφορά την ενεργειακή αγορά έχουμε και κάποιες εξελίξεις που υπονομεύουν την ενεργειακή αγορά. Πρόκειται για τις εθνικές αγορές, την αύξηση της παραγωγής. Αυτό αφορά πολλά κράτη-μέλη Και εσείς τι λέτε, αφού γίνεται τώρα η συζήτηση και η προσπάθεια για μια νέα αγορά, τι θα λέγατε για αυτές τις ε, εθνικές αγορές και την αύξηση των νοοτήτων τους. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας εσείς με όσο είπε η κυρία Χολ, ήθελα να μιλήσω. Και επίση για την αποτελεσματική χρήση της ε, ενέργειας, εκτό από το θέμα της απασχόλησης, να δούμε τι θα γίνει και με την ενεργειακή ταινία. Έχουμε τώρα ένα νέο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα τώρα υπάρχει χρήμα στα διευθυντικά ταμεία για την ενέργεια και η ενεργειακή παινία και στην Ανατολική Ευρώπη σχετίζεται από την κατάσταση των κτηρίων που κληρονομήσατε το παρελθόν. Και, εκεί που μένει ο κόσμος της χώρας της Ευρώπης. Επομένως, εσείς πώς θα μπορούσατε να δώσετε πρόεδρο για όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εντάξετε την, απο... την ε, ε, την, την, αυτή την πολιτική αποτελεσματικότητα στι πολιτικέ που χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία. Τι μπορούσε να είναι το 2014, επίση όσο με την εξωτερική διάσταση. Εσείς προέρχεστε από μία από τις χώρες που έχει μία από τις κορυφαίες ε, εξαρτήσεις μια Οπότε έχουμε κάποια εργοστάσια τα οποία χρησιμεύουν για να εισάγουμε ενέργεια, τα οποία δεν πληρούν όμως τις ευρωπαϊκές προποθέσεις, όπως ας πούμε έχουμε το εργοστάσιο στο Καλίνγκραντ. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα δεν υπάρχει σημείο τόσο ανταγωνισμό, υπάρχει μια ανισότητα. Έχουμε τι δικέ μα εγκαταστάσει με, με τα γνωστά πρότυπα και από την άλλη μεριά εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια τα οποία είναι πολύ πιο κάτω από ε, ε τα δικά μα πρότυπα. Δεν είμαι κατά τη εισαγωγή ε, ηλεκτρική ενέργεια εκτό Ένωση, αλλά θα πρέπει να είμαστε συνεπεί με τα πρότυπα τα οποία τάσουμε. Επίση για την εξωτερική διάσταση. ρίξτε μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία και θα αντιληφθείτε ότι το πρόβλημα που έχουμε για το φυσικό αέριο προέρχεται από το ότι έχουμε κάποιες μακρόπνες συμβάσεις ε, που διέπονται από τη μαθηματική αναπροσαρμογή πάρα πολύ επαχθή. Όπως ας πούμε όλα αυτά τα, τα συμβόλαια με την Ρωσία. Και από την άλλη μεριά βλέπετε πόσο πιο συμφέρουσα σαν ενέργεια είναι αυτό που προέρχεται από το αέριο στη ΣΥΠΑ. Άρα, θυμηθείτε ότι όταν 80% της ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν από, από το, το, τη χρήση του πετρελαίου, τότε κάναμε αυτές τις συμβάσεις με, τη, με αυτή την, ε, α, την πάρα πολύ υπαρχή άτα. Άρα θα πρέπει να κηρυχθεί παράνομη αυτού του είδους η άτα θα καταργηθεί. Θα πρέπει αυτό να είναι κατά τη γνώμη μας ε, πρώτη ερώτηση της Προεδρίας. Ε, pane ministře, já bych teď doporučoval, e, že byste odpověděl na tu první skupinu dotazů, protože byly to dotazy velmi... Αν θέλετε απαντήσετε αυτή την πρώτη ομάδα ερωτήσεων. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. και να μην σας κουράσουν εντός με περισσότερες ερωτήσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ε, πρώτες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιόρταν για την ερώτηση σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας. Αυτή πράγματι είναι μία από τι προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας και προτιθέμεθα να ε, εξετάσουμε το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ελέγξουμε την ε, πρόοδο των ε, κρατών μελών και θα έχουμε μία σειρά συνεδριάσεων θα έχουμε την άτυπη στο Βιλνίους και την επίσημη συνεδρίαση των Υπουργών όπου θα παρουσιάσουμε την έκθεση πρόοδου προς την κοινή αγορά ενέργειας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η στιγμή γιατί μας μένει μόνο ένας χρόνος ε, μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την καταληκτική ημερομηνία. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία περί πυρηνικής ασφάλειας, θέλω να σας πω ότι η Λιθουανική Προεδρία καλωσορίζει ε, την πρώτη πρόταση που κατατέθηκε από την Επιτροπή και προτιθέμεθα να ε, προάγουμε τις ε, συζητήσεις στο Συμβούλιο όσο περισσότερο γίνεται. Και τώρα θα περάσω ε, στην ουσία σχετικά με το τι θα γίνει μετά το 2020. Συγγνώμη, η δική μου ερώτηση για την οδηγία περιπληνικής ασφάλειας ήταν πώς προτιθέ, προτίθεστε να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί επί του θέμα αυτό, αυτού δεν υπάρχουν ε, ε, δυνατότητες ε, συνεργασίας. Η καλύτερη ερώτηση, απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι θα ακούσω την άποψη της Επιτροπής σας. Δεν πρόκειται τόσο για τον συντονισμό. Ε, ξέρετε ότι στο Συμβούλιο ε, συνεργαζόμαστε και εκεί ε, γίνονται και συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα θα πάω στην περίοδο μετά το 2020 όπου νομίζω εκεί πρέπει να αναφέρουμε ότι οι επενδυτές χρειάζονται την προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού πλαισίου και οι αποφάσεις πρέπει να γίνονται υπό υπεύθυνα ε, και σε σχέση ε, με ε, την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να ακούσουμε τα αποτελέσματα από τις δημόσιες διαβουλεύσεις, οι οποίες μόλις ολοκληρώθηκαν. Θα ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις Κομισιόν για τα θέματα αυτά, όπως και προτάσεις ε, σχετικά ε, με συγκεκριμένους τομείς. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση των υποδομών, πράγματι αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά η χρηματοδότηση για ευρωπαϊκά προγράμματα από επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους ε, έτσι ώστε να ε, πολλαπλασιάσουμε τα χρήματα μέσα από εμπορικά προγράμματα. Νομίζω ότι αυτό ε, θα αποτελεί μια σημαντική δυνατότητα να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα για ε, διάφορα προγράμματα τον Νοέμβρη. Θα πάω τώρα στην ερώτηση του κυρίου Πρόντι σχετικά με την αηφορία και τη βιομάζα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, γιατί πράγματι εδώ πρόκειται για μία ερώτηση ε, όπου βρισκόμαστε σε αρκετά αρχική φάση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή ε, εμπλέκει διάφορα κράτη. Και ε, θα αναζητήσουμε την πρόταση της Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρξει και μία συζήτηση ανάμεσα στους αρμόδιους υπουργούς για το θέμα αυτό. Και επίσης πρέπει να ακούσουμε και την άποψη της βιομηχανίας να ακούσουμε ε, τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό ε, το να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Όσον αφορά την ε, ενεργειακή απόδοση, αυτά ετέθησαν από τον κύριο Τούρμες. Μεταξύ άλλων, ε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Και αυτό είναι ένα εργαλείο για να επιτύχουμε τους στόχους μας ε, μέχρι το 2020. Και νομίζω ότι εδώ ε, πρέπει ε, να επικαιροποιήσουμε την κατάσταση γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι βεβαίως και πολύ ενδιαφέρον ε, το να ε, χρησιμοποιεί κανείς ε, την ενέργεια. Όσον αφορά τώρα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, αυτές οι προκλήσεις καταδεικνύουν τη σημασία και τις ευκαιρίες που υπάρχουν πίσω από αυτήν την οδηγία. Όσον αφορά τώρα τα πυρηνικά προγράμματα στη γειτονιά μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Είναι πολύ σημαντική για την ε, περιοχή μας. Και εμείς ε, ανέκαθεν ήμασταν της άποψης ε, ότι τα θέματα ποινικής ασφάλειας δεν σταματάνε στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε λοιπόν να ξέρουμε ότι οι ίδιες προδιαγραφές πρέπει να τηρούνται για να μην αναφερθώ και σε ίσες ευκαιρίες κάτι που είναι πολύ μεγάλη σημασία για ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες διαγωνίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσον αφορά τώρα την ερώτησή σας σχετικά με τη διασύνδεση ανάμεσα σε τιμές αερίου και τιμές πετρελαίου, Νομίζω ότι αυτό ήδη γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή οι μεγάλες ε, ευρωπαϊκές εταιρείες ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση και έχουμε παρατηρήσει ότι αυτή είναι μια τάση που δεν μπορεί να σταματήσει. Και ε, αναμφίβολα ε, θα προσέξουμε, θα βλάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας τις προτάσεις όταν θα εξετάσουμε αυτή τη διάσταση σε επίπεδο υπουργών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ε, ο κύριος Μπούζεκ είναι για να κάνει την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την, για, την για την παρουσίασή σας κύριε Υπουργέ. Είμαι πολύ θερμός οπαδός αυτού του προβλήματος, του προγράμματος του επόμενου εξαμήνου. Κάναμε μεταξύ μας επανειλημμένες συναντήσεις ε, το τελευταίο διάστημα και βεβαίως ε, στο, την περασμένη εβδομάδα η πρόεδρος σας στο Στρασβούργο έκανε μια εξαιρετική ομιλία και πρέπει να πω ότι είστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για το εξάμεινο αυτό. Πιστεύω ότι το επόμενο εξάμεινο θα είναι κρίσιμη σημασία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και μόνο να στηρίξω και να συμφωνήσω μπορώ με τις ερωτήσεις των συναδέλφων και τις ε, δικές σας απαντήσεις. Θέλω να προσθέσω κάτι στο ζήτημα της, ε, της υποδομής που έθεσε η κυρία Γιόρντον λόγω των, ε, των, των θεμάτων που έχουν σχέση με τα έργα που έχουν κοινοτικό ενδιαφέρον για να σταματήσουμε και τα ενεργειακά νησιά. Ε, ε, η ερώτηση επίσης του συναδέλφου Τούρμες είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή η, σύνδεση της τιμής του, ε, του αερίου με τον πληθωρισμό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, αν λάβουμε κυρίω υπόψη μα τη διαφορά τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε σχέση με τι ΗΠΑ. Και ένα άλλο ζήτημα. Θα πρέπει το, να επιτρέψουμε το διαμεθοριακό ενεργειακό εμπόριο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν έχουμε κωδικού ε, χρειάζομαστε κώδικες μεταβίβασης και, άλλα, και άλλες προϋποθέσεις. Αλλά το δυσκολότερο ίσως να είναι η συμβατότητα των προγραμμάτων στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν για να επιτευχθούν ε, σωστά καλά αποτελέσματα για να δημιουργήσουμε, ένα άλλο ζήτημα επίσης είναι η δημιουργία μιας αγοράς ε, φιλικής προς το χρήστη. Πώς θα ε, ε, υλοποιήσουμε, πώς θα εκμεταλλευτούμε τα επιτεύγματα της πληροφορικής, πώς θα μπορέσουμε πραγματικά να το κάνουμε αυτό εύκολο για τους πολίτες μας, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς γίνεται στην αγορά και πώς θα μπορέσουμε να τους ε, επιτρέψουμε να έχουν την σωστή επιλογή στο θέμα της παροχής ενέργειας, πώς θα τους βοηθήσουμε να αποφασίσουν μέσω των τοπικών ενδιάμεσων, κάτι που επίσης είναι εφικτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση, ο κ. Πέντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω... Ευχαριστώ πολύ που παρουσιάσατε το πρόγραμμα αυτό και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη από το 2014 χρειάζεται μια εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε όμως μια διαφανή σταθερή αγορά. Ε, και ε, όταν ε, πρόκειται για ε, σταθερές ε, και διαφανείς αγορές υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ε, λέμε ότι στην αγορά ενέργειας θα πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, όμως Κάποιες χώρες πληρώνουν για αέριο από την Gazprom διπλάσιες τιμές από ότι η Γερμανία. Έχω την αίσθηση ότι οι συνάδελφοι στη Βαλτική αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και όσον αφορά την αηφορία ε, σχετικά με τους ε, στόχους αηφορίας αλλά και δεσμευτικούς στόχους ε, γιατί δεν γίνεται λόγος για το ότι Μπορεί κανείς να περιορίσει τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Και οι χώρες της ε, Βαλτικής ε, για πόσο καιρό ακόμα θα πληρώνουν διπλάσια από τη Γερμανία και τι μπορεί να κάνει ο κύριος Υπουργός έτσι ώστε οι επενδυτές να μπορούν να γνωρίζουν τι θα γίνει μετά το 2020. Γιατί το 2020 είναι πολύ κοντά ε, για τις, ε, για πολλές επιχειρήσεις ε, και πρέπει να ξέρουμε, οι επιχειρηματίες πρέπει να ξέρουν τι είναι προβλέψιμο για αυτούς. Τελευταία ερώτηση αυτή από μέλος της Επιτροπής, οπότε αν θέλετε απαντήστε σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στον κύριο Πούζακ. απαντήσω πρώτα. Η επιλογή, η διαδικασία επιλογής των PCI, των έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος, είναι πολύ σοβαρή, έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση και αυτή την εβδομάδα που γίνονται κάποιες προκαταρτικές συζητήσεις για τον κατάλογο των έργων με κοινοτικό ενδιαφέρον που θα οριστικοποιηθεί. Προσβλέπουμε στο, στην, στην οριστικοποίηση το φθινόπωρο όπως σας είπα. Θα δώσουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην διάσκεψή μας στα έργα κοινού ενδιαφέροντος. Χαίρομαι πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και να παρουσιάσετε και την έκθεσή σας. Αυτό για μας αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο ε, προς τα κράτη-μέλη για να δώσουν ε, προσοχή στα όσα έχει να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού. Τα προγράμματα, η συμβατότητα των προγραμμάτων στήριξης. Περιμένουμε κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα αυτό και σε προσβλέπουμε ένα, σε ένα μηχανισμό συνεργασίας που θα υποβληθεί φέτος το καλοκαίρι. Κατόπιν θα παρουσιαστεί αυτό και θα συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο. Διότι πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντικό στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης το πώς δηλαδή θα πρέπει να λειτουργήσει η κοινή αγορά και το πώς θα πρέπει να αποφύγουμε να είναι αντιφατικά μεταξύ τους τα διάφορα προγράμματα στήριξης του κάθε κράτους μέλους. Ας περάσω τώρα στα ερωτήματα του κυρίου Μπέντσεν. Πράγματι η διαφάνεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ότι η φυστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει ε, όλο και περισσότερη διαφάνεια. Είμαι πεπισμένος ότι μετά την πλήρη υλοποίηση ιδίω του τρίτου ενεργειακού πακέτου με τις απαιτήσεις του θα έχουμε ανεξάρτητους ε, παρόχους ε, ενέργειας και αυτό θα αυξήσει τη διαφάνεια. Όπως επίσης θα υπάρξει και πολύ μεγαλύτερη διαφοροποίηση, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί είναι οι άλλοι πυλώνες, τους οποίους μπορώ να αναφερθώ, για το τι θα πρέπει να γίνει, το τι γίνεται ε, και σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχουν και τα νομικά μέσα, αλλά και η διαφοροποίηση και οι εναλλακτικέ οδοί ε, προμήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, εκ μέρου όλων των συναδέλφων. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τις ε, πολύ σαφείς απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε επίσης για όλα όσα μας είπατε. Αποτελεί για μας ε, μεγάλη τιμή που ήρθατε ήδη από την αρχή στη δική μας Επιτροπή, γιατί πράγματι η ενέργεια αποτελεί ε, μία από τις βασικότερες προτεραιότητες των εργασιών μας. Ε, ήδη χαιρόμαστε που θα σας ξανασυναντήσουμε στην Επιτροπή μας. Έχουμε πλήρη συνέστηση ότι η ενέργεια και όλα τα σχετικά με αυτήν αποτελούν ένα κρίσιμο θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, για όλα τα κράτη-μέλη και τους πολίτες της. Είναι θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε και βεβαίως ευχόμαστε μεγάλη επιτυχία στην, στο έργο σας στην Λιθουανική Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Bene, allora proseguiamo. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν τις ε, εργασίες μας ε, αφού ακούσαμε τον ε, νεότατο Υπουργό και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Πιλάρ που θα μας μιλήσει για το υπολογιστικό νέφος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σήμερα για πρώτη φορά να συζητήσουμε την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία, η οποία αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το νέο τη πληροφορική. Όπω γνωρίζετε, εδώ θα διαμορφώνει τη θέση του Κοινοβουλίου κατά με τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει επίση να μην ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια βασική δράση για την ψηφιακή ατζέντα τη επιτροπή. Και αυτό το φαινόμενο το ονομαζόμενο υπολογιστικό νέφος είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας. Και Έχουμε διάφορους μεταβλητές που δημιουργούν ένα περιβάλλον πάρα πολύ εξαιρετικής υφής. Πρόκειται για έναν χώρο που δεν συνδέεται με βάση δεδομένων ούτε με δίκτυο. Η ιδέα είναι χρήστες, μπορεί να είναι επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα ή θεσμικά όργανα και σε πάρα πολύ λίγα χρόνια θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι αυτό το cloud ε, είναι κάτι που δημιουργεί πάρα πολλές υποσχέσεις γιατί πρόκειται για έναν ε, κλάδο όπου αναπτύσσεται ε, πιο γρήγορα από όλους όσον αφορά την επικοινωνία. Για να μην πούμε ο πιο μεγάλος, ο τομέας με την πιο γρήγορη ανάπτυξη. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι χρειάζονται εδώ πέρα κάποιες εφαρμογές, κάποιες ε, υποδομές, θα πρέπει η, αντίδραση, η λειτουργία να είναι σχεδόν ε, κεραυνοβόλα. Οπότε αυτό έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο όλες οι επιχειρήσεις έχουν συλλάβει το πόσο σημαντικό είναι το νέφος και την παραγωγικότητά τους. Πρόκειται για κάτι το οποίο δίνει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Δεν θα υπησέλθω σε όλες τις ε, λεπτομέρειες, τις θετικές, σε όλα τα καλά, τα πλεονεκτήματα που προσδίδει αυτή η ε, τεχνολογική εξέλιξη. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εύστοχα τα λέει στην παρουσίασή και έχει εντοπίσει τρεις διαφορετικούς τομείς όπου θα πρέπει να μείνουμε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμβάλλει ε, σε κάποια σημεία και ανέλαβα και εγώ την έκθεση για αυτό το λόγο για να συμπληρώσουμε τόσο έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πέντε, σε πέντε τομείς. Σε πέντε τομείς που θα πρέπει να χαράξουν μια σωστή στρατηγική για το νέφος οπότε και μετά η Ευρώπη μπορεί σε σχέση με το νέφος να βοηθήσει ε, και για την απασχόληση και για την οικονομική ανάπτυξη. Πρώτα πρώτα. Πρόκειται. Για το δυναμικό του πολιτιστικού νεύους. Σε το γύρο ότι ε, συμμετέχουμε κατά 24%. Και σύμφωνα με την έκθεση της κινητικότητας χρειαζόμαστε για την ε, πληροφορική 700 με 1 εκατομμύριο ε, ειδικού. Άρα και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες δράσεις μελέτης, ενασχόλησης με το δυναμικό αυτού του νέφους. Δεύτερος τομέας αφορά την ασφάλεια σε σχέση με το νέφος και επίσης το ότι θα πρέπει να υπάρχουν θεμητές συνθήκες ε, ανάπτυξης στο νέφος. Χρειάζεται επίσης να σκεφτούμε ότι μας και επίσης η οδηγία για τις υπηρεσίε πρόκειται να συμβάλλουν. Επίσης όσον αφορά τον ε, ε, δημόσιο τομέα. Είναι πολύ σημαντικό το νέφος γιατί και ο το τομέας έχει μεγάλη σημασία ε, στις οικονομίες μας. Οπότε οι δυνατότητες του νέφους που μας οδηγεί σε πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου αυτό σημαίνει όφελος για όλους τους πολίτες. Υγεία, κινητικότητα, αποτελεσματικότητα, παιδεία και επίσης λιγότερο κόστος για τις ε, επιχειρήσεις. Αλλά πέραν αυτών, ακριβώς επειδή το δημόσιο έχει τέτοιες στην Ευρώπη, εάν μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη του νέφους, τότε θα έχουμε το φαινόμενο της μόχλευσης. Για πολλούς οικονομικούς τομείς, τομείς οικονομικής δραστηριότητας και του ιδιωτικού τομέα. Άρα θα είναι σοβαρέ επιπτώσει του νεύου. Και μιλάμε για την πληροφορική που τώρα δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ στο δημόσιο και στι υπηρεσίε του. Άρα θα πρέπει να αγκαλιάσει το δημόσιο το νέφος, το υπολογιστικό. Άρα και πρέπει να επιταχυνθεί η πορεία προς την εταιρική σχέση για την ε, ανάπτυξη του νέφους του υπολογιστικού. ακριβώ, όπως προτείνει το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, τα ταυτοστομία είναι τα πρότυπα τα οποία διέπουν το υπολογιστικό νέφος να αποφύγουμε μία αγορά όπου οι χρήστες είναι όμοιροι, εχμάλωτοι ενός παρόχου. Άρα χρειάζεται να είναι ε, εύκολη, ευέλικτη η φορητότητα και να υπάρχει λειτουργικότητα ούτω ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον η φορητότητα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε μια καταγραφή των προτύπων και μέχρι τις 4 ε, ενάτου με τις τροπολογίες θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλα αυτά τα οποία ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσης θα ωφεληθούν από πλευράς διαφάνειας και ενημέρωσης οι καταναλωτές από το νεφος. Επίσης, κάτι το οποίο κατάλαβα από τις που έκανε για αυτό το θέμα, οι επιπτώσεις μιας ε, εύστοχης στρατηγικής για την ανάπτυξη του πολιτισμού νεύου στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει απομονωμένα, μόνο εδώ στην Ευρώπη, σε απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συνεργασία με άλλες περιοχές του κόσμου. Ε, και βεβαίως θα πρέπει να συνοηθούμε και να ενεργήσουμε από κοινού με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά θα πρέπει να δούμε το πώς θα αναπτύξουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά. Και έτσι να δοθεί όθηση στην ε, τόσο καταπλημένη αυτή αγορά. Αυτά. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τώρα ε, τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την ε, τελευταία εβδομάδα πριν από τις θερινές διακοπές. Οτιδήποτε προτάσει έχουν οι συνάδελφοι, ερωτήσει, Πρέπει να απαντήσω. Έχουμε το Σεπτέμβριο μια ανάγνωση, μια πρώτη συζήτηση. Οπότε στα πλαίσια αυτής της ε, συμβολή μου για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω να πω το ότι νομίζω πω το κοινό μπορεί να βοηθήσει και σημαντικά τίποτε άλλο. Πιλάρ, σε ευχαριστώ. Κύριε Κάλφιν, που θα αντικαταστήσετε κάποια συνάδελφο που δεν μπορεί να παραστεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη και μάρες του συναδέλφου μου. Θέλω να εκφράσω τις απόψεις του σκιώδους συγητή της Σοσιαλιστικής Ομάδας για την έκθεση για το υπολογιστικό νέφος. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Τεκαστήγιο για την εκτεταμένη σε βάθος ολοκληρωμένη έκθεση η οποία επισημαίνει τις βασικές δυσκολίες ε, του υπολογιστικού νέφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις του σκανδάλου Prism και χωρίς βεβαίως αυτό να επηρεάζει τις ε, ε, αρμοδιότητες των άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου, υπό την επιφύλαξη αυτών των αρμοδιοτήτων, θέλω να επισημάνω ότι εκτιμά την σημασία ε, των, ε, του υπολογιστικού νέφου στην ευρωπαϊκή στρατηγική και η έκθεση αυτή με τους πυλώνες νομίζω έρχεται στο να θίξει τις και είναι πολύ σχετική με τις πρόσφατες εξελίξεις. Ε, κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα του, ε, της έκθεσης. Πρώτον, η σχετική υποδομή. Ε, καταρχήν, υπολογιστικό νέφος σημαίνει ότι για να χρησιμοποιηθεί αυτό σωστά χρειάζεται σωστά, σωστές ευρυζωνικές συνδάσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε την προσπάθεια να έρθει η ευρυζωνικότητα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κυρίως θα αποτελέσει δυσκολία και για τα άτομα αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κυρίως αυτές που βρίσκονται σε κάπως αραιοκατοικημένες περιοχές που έχουν χαμηλότερη πρόσβαση τις ε, βριζονικές συνδέσεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για το θέμα του υπολογιστικού νέφους θα πρέπει αναπόφευτα να θέσουμε ε, και το θέμα του ψηφιακού χάσματος αλλά και ε, τη δυνατότητα να, να βαθυνθεί αυτό έτσι περαιτέρω. Επίσης, όταν μιλάμε για υποδομές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι προς το παρόν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έλλειψη ε, σερβερ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σχέση και αυτό με το σκάνδαλο. Ε, όταν μιλάμε για νέφος είναι δύσκολο να το εντοπίσουμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να αναπτύξει αυτή την υποδομή για να βρίσκεται σε ίση βάση με στον υπόλοιπο κόσμο. Όσον αφορά τις δεξιότητες τώρα και αυτό το επεσήμανε η Πιλάρ ε, και εκ μέρους της Κατρίν Τρότμαν θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω τις, ε, τα ευρήματα αυτά. Όχι μόνο χρειαζόμαστε περισσότερη εκπαίδευση για τους χρήστες, αλλά περισσότερα προγράμματα προσόντων για την ειδική διαχείριση του υπολογιστικού νέφους και την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής αυτής. Από, την κοινωνική, από κοινωνική σκοπιά τώρα θα πρέπει επίσης να παρακολουθούμε όταν αναπτύσσουμε το υπολογιστικό νέφος και τη σχετική υποδομή να παρακολουθούμε τις επιπτώσεις του ε, στο, ε, στην κοινωνία. Ας πούμε την απόσταση μεταξύ των ειδικών ε, πληροφορικής και άλλων ειδικών στις επιχειρήσεις, το γεγονός ότι οι διάφορες συμβάσεις μπορεί να υπονομεύσουν την καινοτομία και την βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ε, έχει να, να δοθεί έμφαση στο θέμα της καινοτομία. Επίσης πρέπει η φορητότητα και η διαλειτουργικότητα να ενθαρρυνθούν όπως είπε και η Πιλάρ. Τώρα, αυτό το οποίο σαφώς εμείς πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να μην αναφερόμαστε στην, ανάμεσα στις διαφορές των εθνικών στρατηγικών υπολογιστικού νέφους, αλλά να διακρίνουμε ανάμεσα στις, στην ευρωπαϊκή και τη μη ευρωπαϊκή στρατηγική. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος, να μπορεί αυτός να συγκρίνεται με τις εξωτερικές αγορές και να περιορίζονται οι, πιθανώς οι διαφορές με στο εξωτερικό. Επίσης, η στρατηγική που θα ξεκινήσει από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει ένα διεθνές σκέλος και θα πρέπει να συνδέεται με οποιασδήποτε προσπάθειες γίνονται εκτός Ένωσης για την ανάπτυξη προτύπων και οι, δυνα, οι δυνατότητες αυτές στο, τομέα του υπολογιστικού νεύου θα πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερα. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι η παράγραφος 4 ίσως είναι εξαιρετικά ουδέτερη ε, γιατί λέει ότι δεν θα πρέπει να δοθεί πλεονέκτημα σε κανένα ε, επιχειρηματικό μοντέλο. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ε, την ε, ομιλία του Αντιπροέδρου στον Ταβός, του Ταλικρού στον Ταβός, είπε ότι θέλουμε όχι μόνο να, έχουμε φιλικότητα προς τον νέφος, αλλά να έχουμε και δραστηριότητα ε, σε σχέση με τον νέφος, δηλαδή να είμαστε παραγωγικοί και να προσφέρουμε ε, εμεί λύσεις και όχι απλώς να χρησιμοποιούμε λύσεις που έχουν αναπτυχθεί κάπου αλλού. Καλό λοιπόν ε, να προωθηθούν τα, ε, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ζητήσω ε, συγγνώμη του που σας άφησα και ε, λιγάκι παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Συνάδελφο Ρόντε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την, το σχέδιο της έκθεσης από την Πιλάρ που κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ καλό και εξετάζει όλες τις ε, ενέργειες ε, που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, στους φιλεύθερους εμείς ε, συμφωνούμε με αυτό που ελέγχει σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το υπολογιστικό νέφος έτσι ώστε να είναι πράγματι πιο αποτελεσματικές οι δημόσιες υπηρεσίες ε, και να είναι πιο αξιόπιστες και οι ηλεκτρονικές προμήθειες. Επίσης ε, πρέπει να προσφέρεται η ασφάλεια, η αξιοπιστία, οι πληροφορίες ε, να μην διατίθενται σε όλους αλλά σε έναν ορισμένο αριθμό ενδιαφερόμενων. Και εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να είναι ουδέτερη και ανοιχτή σε όλους τους παρόχους υπολογιστικού νέφους ε, και όλοι να είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο. Όσον αφορά τις ε, προδιαγραφές ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προηγηθεί και τέλος οι φιλελεύθεροι στηρίζουν αυτό που αναφέρεται σχετικά με την προστασία του καταναλωτή. Με την έννοια ότι οι καταναλωτές πρέπει και αυτοί να έχουν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ε, πριν τελικά ε, καταφύγουν και αυτοί στο υπολογιστικό νέφος και χαίρομαι, προσβλέπω στη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ ε, αντεστότε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Ε, την έκθεση της Κομισιόν τη βρήκα στην αρχή λιγάκι παραπλανητική. Μου δημιούργησε έτσι μια σύγχυση γιατί υπάρχουν ε, πάρα πολλές εκδοχές. Το Eurocloud, η Κομισιόν επίσης ε, ξέρει ότι και χρηματοδοτεί αυτά σε αρχική φάση και διερωτήθηκα γιατί τα αναφέρει τώρα η Κομισιόν και όχι παλαιότερα ή γιατί δεν περίμενε να υπάρξει κάποια τάξη στο υπολογιστικό ε, νέφος στην Ευρώπη. Η κυρία Ντεκαστήγιο νεφο στην ευρωπη η ότι θα βοηθήσει στο να υπάρξει κάποια τάξη. Τα πέντε σημεία που αναφέρει είναι ε, με σωστή τάξη και ε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προδιαγραφές, τη διαφάνεια ε, να υπάρχει κάποια καθοδήγηση σε αυτό τον τομέα. Επίσης, ε, συμφωνούμε με τις επιφυλάξεις της κυρίας Τράουτμαν για την κοινωνική πτυχή του υπολογιστικού νέφους και ίσως αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε περισσότερο. Πολλά από τα μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιγράφονται ως ε, πλασματικά. Πολύ λίγοι έχουν τον πραγματικό έλεγχο. Και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι πολίτες ε, πολλές φορές ε, ε, βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο, είναι οι μικροί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους μεγάλους και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά τοποθετώντας την στρατηγική αυτή σε ένα σωστό πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι η έννοια της ε, ε, φορητότητας των ε, δεδομένων είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή και όλους τους άλλους σκιώδεις γιατί νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε παραγωγικές συζητήσεις και χαίρομαι πολύ που έχουμε έτσι ένα πολύ καλό σχέδιο για να ξεκινήσουμε με αυτό ως βάση. Το Ζανόφσκι παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Συμφωνώ με όσου είπα καλά λόγια για την έκθεση της συναδέλφου. Πάρα πολύ πλήρης αυτή η έκθεση. Εξηγεί πάρα πολύ καλά τη φάση την οποία έχουμε φτάσει όσον αφορά την εξέλιξη αυτού του νέου Επίση εξηγεί και το όραμα που έχουμε για το μέλλον και μέσα σε λίγες ε, σελίδες περιγράφεται μια πάρα πολύ περίπλοκη πορεία. Ακόμη και οι ειδικοί στην πληροφορική πάντοτε δεν μπορούν να συλλάβουν όλες τις λεπτομέρειες αυτού του φαινομένου. Ε, και νομίζω ότι ήρθε σε σωστή στιγμή αυτή η έκθεση ε, γιατί συζητούμε πάρα πολλέ εκθέσεις και ε, επίσης με αυτές τις εκθέσεις ε, Ιδίω όσον αφορά την, την έκθεση Ρόντα για την ε, ψηφιακή ατζέντα, τα πράγματα, η εξέλιξη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Επίση, θα πρέπει να βροντίσει η Ευρώπη την, ε, την ψηφιακή υποδομή, αλλά πάλι η χρήση του νέφους της πληροφορικής θα βοηθήσει πάρα πολύ ε, θα συνδυαστεί με άλλες τεχνολογικές πρόοδου όπως την ευρυζωνικότητα και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διακινούμε ε, τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Γιατί βλέπουμε ότι σήμερα ε, επιβάλλεται η διαβίβαση πάρα πάρα πολλών δεδομένων. Πάρα πολλοί συναδελφοί επίσης ανέφεραν την συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό και επίσης αναφέρθηκαν οι διάφορες παράμετροι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όσον αφορά ε, την διείσδυση του ιδιωτικού στο δημόσιο τομέα και επίσης όσον αφορά τις διοικητικές παρεμβάσεις. Προσοχή να μην φρενάρουμε ε, αυτή την εξέλιξη. προσοχή να λάβουμε υπόψη την εμπειρία κάποιων χωρών όπου η γραφειοκρατία σταμάτησε την εξέλιξη. Επίσης, όπως είπαμε και πρέπει να λάβουμε υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων και να δούμε πώς θα γίνει ο χειρισμός, ε, η διαχείριση αυτού του πολιτικού νέφους με ασφάλεια θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες σχετικώς. Επίσης θα υπάρξει περισσότερη ενημέρωση του κόσμου σε σχέση με την διαβίωση των δεδομένων. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει νέφος πληροφορικής. Πρέπει να υπάρχει ε, ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον έλεγχο βουλευάς ε, διοίκησης. Πιστεύω σε αυτή την έκθεση και θα συμβάλλω τα μέγιστα ώστε να επιτυχεί τις προσπάθειες της εισηγήτρια. Ευχαριστούμε κύριε Τόσενόφης κύριε Πρόεδρε. Έχει το λόγο κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ ε, Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον, τη συνάδελφο Καστίγιο για την έκθεσή της. Ε, το υπολογιστικό νέφος ε, υπόσχεται πάρα πολλά, είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο γιατί προσφέρει πάρα πολλές προοπτικές κυρίως στο να μπορεί να συγκρατήσει, έχει πολύ μεγάλη μνήμη ε, και πολύ καλές δυνατότητες υπολογισμού, κάτι που ε, είναι αντίθετο να το σκεφτεί κανείς ε, σε σχέση με μεμονωμένους χρήστες. Άρα δηλαδή, εδώ έχουμε μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε το υπολογιστικό νέφος ευρύτερα, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια, κυρίως όσον αφορά τα δεδομένα, ε, να μην είναι αντικείμενο ε, δόλιων χειρισμών. Και επίσης, και να μην μπορεί να υπάρξει κατασκοπία, να μην χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα με τρόπο που κρίνεται κατάλληλος. Πέρα λοιπόν από, αυτό το, από αυτή τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί, νομίζω θα πρέπει να αξιολογήσουμε με πολλές περισσότερες λεπτομέρειες τους κινδύνους που υφίστανται, τόσο για την διαθεσιμότητα των δεδομένων, όσο και για το ότι τα δεδομένα ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, ενδεχομένως για διαφορετικούς σκοπούς. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγγύησεις πριν τελικά ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ε, κάποια συγκεκριμένη στιγμή ενδεχομένως να μην μπορούμε καν να το ελέγξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς η Αντζέλικα, Αγγέλικα μάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστώ θερμά την εισηγήτριά μας για αυτή τη θαυμάσια έκθεση, το σχέδιο της έκθεσής της. Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στην έκθεση αυτή που μπορούμε να τα δούμε με την ησυχία μας. Ορισμένοι συνάδελφοι τα έθιξαν ήδη. Ε, κατά την τελευταία συνεδρίαση είχαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις υποκλοπές, το τι θα κάνουμε ως Ευρωπαίοι και ε, από τον πρόεδρο της Εστονίας αναφέρθηκε ότι θα πρέπει πράγματι να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό cloud ε, το θέμα είναι βέβαια τι σημαίνει αυτό, τι, πώς το ερμηνεύουμε ο καθένας μας και πού ξεκινάμε. Ε, νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσουμε και εμείς τη δική μας την έκθεση πριν καταθέσει δική της έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα στην έκθεση δικαστήριο είναι ότι σε όλη την έκθεση αναφέρεται σε θέματα εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη κυρίως όσον αφορά την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ε, σε όλους ότι ε, τα δεδομένα τους είναι προστατευμένα, τότε νομίζω δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να ε, δημιουργήσουμε, να προκαλέσουμε εμπιστοσύνη έτσι ώστε να βρούμε ένα ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος. Όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, υπάρχουν στην έκθεση ε, και νομίζω ότι ε, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε προς ένα ευρωπαϊκό λογιστικό νέφος. Θα πρέπει, αν θέλουμε να υπάρχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τότε θα πρέπει να έχουμε ε, ένα ελάχιστο όριο προδιαγραφών να μπορεί κανείς να τις επικαλεστεί. Από πλευράς προσέγγιση, όλα αυτά βρίσκω πολύ σημαντικά, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η πολιτική συζήτηση. Ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούμε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ε, υπολογιστικό νέφος και αυτό που με σοκάρει είναι οι εξελίξεις ε, τις οποίες παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, ε, εμείς ε, στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό ε, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι. Δηλαδή ένα ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος σημαίνει ότι κέντρα δεδομένων θα πρέπει να υπάρχουν μόνο στην Ευρώπη. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος σημαίνει αυτό ότι ε, τη μεταφορά θα μπορούμε να την ε, επιτρέπουμε και σε άλλες περιοχές του κόσμου ή επίσης συγκεκριμένα τελικά τι θα κάνουμε με τη συμφωνία που έχουμε συνάψει με τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως αυτά θα πρέπει να τα διαπραγματευτούμε εκ νέου. Υπάρχει εδώ μια σειρά θεμάτων και νομίζω ότι η δική μας Επιτροπή είναι εκείνη που πρέπει να τοποθετηθεί. Αυτό που μου λείπει λιγάκι είναι ότι δεν έχω έτσι ακριβώς μια ε, συγκεκριμένη εικόνα. Ε, συζητάμε εδώ και μισή ώρα ε, για το θέμα των ε, ιδιωτικών τελών, πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε όλα αυτά και κατά πόσο ενδεχομένως χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και όλα αυτά σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Υπολογιστικό Νέφος. Επαναλαμβάνω πού ακριβώς θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και τι ακριβώς είναι απαραίτητο για να μπορούμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Υπολογιστικό Νέφος είναι καθοριστική σημασία για τους πολίτες μας και τις επιχειρήσεις μας. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που είναι ανοιχτά και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τη συνάδελφο. Bene, abbiamo terminato. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν τις ε, παρεμβάσεις και τώρα ε, θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θέλω καταρχήν να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ε, υποβάλει κάποια σχόλια εν ώψη της γνωμοδότησης. Θέλω λίγα πράγματα μόνο να προσθέσω πέραν αυτών. Ε, είμαστε πολύ υπέρ της ανάπτυξης των ευρυζωνικών συνδέσεων. Είναι πολύ σημαντικά για το υπολογιστικό νέφος. Τώρα όσον αφορά το θέμα των υποδομών. Θέλω να καταρχήν να πω ότι αυτός δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφευθεί ο κίνδυνος πρόσβασης στα δεδομένα από ξένες κυβερνήσεις. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη ε, online. Χρειάζεται ένα διαφανές πλαίσιο, χρειάζεται ε, χορηγία, ενίσχυση της ευρείας έρευνας και πρέπει επίσης να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους οι ξένες κυβερνήσεις να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Το δεύτερο τώρα. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στην υποδομή της Ευρώπης. Να σκεφτούμε τη δυνατότητα όπου σε μια περίπτωση που θα υπάρχουν ε, κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη να υπάρχει δυνατότητα κάποιες υπηρεσίες να παρέχονται από αμερικανικές επιχειρήσεις. Μην ξεχνάμε ότι ε, ε, υπάρχουν και εφαρμογές που είναι εξωχωρικές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από εξωτερικές ε, εταιρείες. Αυτό δεν αρκεί για να πούμε ότι τα δεδομένα αυτά, στα δεδομένα αυτά έχουν πρόσβαση ξένες κυβερνήσεις. Όσον αφορά τη γνωμοδότηση, θέλω να πω κάτι ε, σχετικά με την προστασία του καταναλωτή. Το γεγονός ότι της χρήσης του υπολογιστικού νέφους. Θέλω να επαναλάβω εδώ ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι οι υπηρεσίες του νέφους στο μέλλον θα χρησιμοποιούνται παντού. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς όπως και το διαδίκτυο. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν μπορεί κανείς να συγκρίνει αυτού του είδους τις υπηρεσίες με τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Το να πει κανείς λοιπόν ότι θα χρησιμοποιούμε το υπολογιστικό νέφος ως βασικό ως βασική μέθοδος θα είναι σαν να λέμε ότι και το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως βασικό μέσο. Και επίσης οι πελάτες δεν αναγνωρίζουν, δεν διακρίνουν αυτά τα δύο. Λοιπόν, πρέπει και αυτοί να έχουν τη γνώση ότι θα χρησιμοποιήσουν ή δεν θα χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες νέφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απολύτως βεβαία ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει διατυπωθεί αυτή η πρόταση, η γνωμοδότηση μάλλον ε, ε, και η προσέγγιση του θέματος του καταναλωτή είναι σωστό. Αυτό έχει ισχύσει στο παρελθόν και με τον κανονισμό για τα cookies και ίσως ε, να γίνει μια ανακοίνωση για τους όρους των πρότυπων συμβολέων που κατά κάποιο τρόπο θα αυξήσουν την ε, προστασία του καταναλωτή. Θέλω να αναφερθώ επίσης και στα δικαιώματα, ε, τα πνευματικά δικαιώματα. Χαιρόμαστε που η πρότασή μας, η σύστασή μας έχει ληφθεί υπόψη όσον αφορά την επιβολή τελών, ιδιωτικών τελών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στον τομέα του υπολογιστικού νέφους. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του τομέα αυτού και θεωρούμε ότι το θέμα του υπολογιστικού νέφους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Να σχολιάσω επίσης και τη διαφορά μεταξύ στρατηγικής Ευρώπης και στρατηγικής εκτός Ευρώπης. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια εταιρική σχέση. Ε, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Παρότι τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν δική του στρατηγική υπολογιστικού νέφους, η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση βοηθά στην ανταλλαγή ιδεών μεταξύ χωρών και εμπειριών βεβαίως μεταξύ χωρών. Υπό την έννοια αυτή πιστεύω ότι προσπαθούμε να πετύχουμε μια ευρωπαϊκή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιλάρ, τα συμπεράσματά σου. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την τόσο θετική τους ε, αξιολόγηση του σχεδίου κειμένου. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις της. Θα υπάρξει ο χρόνος μετά τι περινές διακοπές, αρχές Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να συνδεθούμε και οδησίγητες ούτως ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία που να καταλήξει στην Ολομέλεια τέλος του έτους. Και επίσης ανέφερες, ε, αναφέρθηκαν μάλλον πάρα πολλά σημεία. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλα. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Άρα ραντεβού το Σεπτέμβριο. Grazie Pilar, grazie a tutti i colleghi. Pilar, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους που έλαβαν τον λόγο και σας πενθυμίζω ότι η καταληκτική πρόθεσμη για τι τροπολογίε είναι η Τετάρτη 9 το μεσημέρι. 14 Δεκάτου ε, θα ψηφιστεί η έκθεση στην Επιτροπή και το Νοέμβριο, το Νοέμβριο στην Ολομέλεια. Και τώρα η κυρία Βαλεάν δεν είναι εδώ. Την αντικαθιστά ε, ο συνάδελφος ή συνάδελφος ή συνάδελφος Χολ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα αντικαταστήσω την κυρία Βαλιάν. Λέει κυρία Χολ. Να σας διαβάσω μια δήλωση την οποία συνέταξε για το θέμα. Λέει, αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως διαγνωστεί ότι ο εν λόγω κανονισμός Όσο αφορά την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Παιδευτικών Σχεδίων, συνεργειακή υποδομή εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ΙΔΙΑ έχει υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009. Τότε δε η κυρία Βαλιάν επίση ήταν συγγετρία τη Ίτρε και σε συνεργασία, σε με την ε, Γιούρη, αποφασίστηκε να προσφύγουμε κατά του Συμβουλίου για την ε, νομική βάση και έτσι αμφισβητήσαμε τον ε, κανονισμό. Και έχουμε επομένω το άρθρο 337 που επικαλεστήκαμε και το, το 187. Αυτή ήταν η νομική βάση, είπε το Συμβούλιο. 337 και 187. Γιατί αφορούν τη δραστηριότητα ε, συλλογή ε, γενικών πληροφοριών. Και είπε τότε, κύριε Βαλιάν, ότι αυτό ο οργανισμό δεν αφορά μόνο τη συλλογή πληροφοριών, αλλά διαμορφώνει την μέλουσα πολιτική ε, της ενέργειας γιατί έτσι δημιουργείται μια πλήρη εικόνα για την υποδομή. Και σύμφωνα με την συνθήκη αγώνας για την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου στην ενεργειακή πολιτική, ε, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να προβλέπεται στην απόφαση Όντω, έκρινε στις 6 Ιανουαρίου του 2012 το δικαστήριο ότι πρέπει να ακυρωθεί ο λογοκονισμός και ότι θα πρέπει να προτείνει σε νέα νομική βάση. Ε, την, ε, μια καινούργια πρόταση τέλο και με συναπόφαση να, συ, να κρίνει το Κοινοβούλιο. Και είπαμε ότι επίση ότι αυτή η πρόταση είναι ίδια με τον οργανισμό, αλλά όμω παρά πολλέ τροπολογίε του Κοινοβουλίου, η κυρία Βαλιάν του 2010, έλειψαν υπόψη από την ε, Επιτροπή. Ο δε κανονισμό απαιτεί το ότι μέσα σε δύο χρόνια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν όσον αφορά τα εμβλητικά προγράμματα για κατασκευή, εξυγχρονισμό ή κλείσιμο σταθμών ε, δημιουργία ε, παραγωγή ενέργεια. Και αυτό να αφορά και τι ε, τις του εξουδίου του Άδραγα και από ο κανονισμός είπε ότι θα πρέπει να κοινοποιούνται στα, και στα κρατημέλη όσα δεδομένα χρειάζονται. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επομένως προχώρησε σε μια τέτοια κοινοποίηση. Οπότε με όλα τα δεδομένα τα οποία μπορούν να συλλεχθούν μπορούμε τώρα να εντοπίσουμε το τι προβλήματα υπάρχουν σε ζήτηση και προσφορά για την ενέργεια. Χρειάζεται ένας τέτοιος ε, κανονισμός, θεωρεί συγκίτρια, και για την ε, ε, Connecting Europe Facility. Οπότε να συμπληρωθεί το έργο που γίνεται στην ειδική υποδομή, να έχουμε ασφάλεια της προσφοράς και να συνδέονται στο γενικό δίκτυο η ενεργειακοί πόροι. Θέλω κύριε Βαλέαν και έχουμε αυτήν τώρα την έκθεση και με κάποιες τροπολογίες, ξεράζω κάποιες έννοιες, πρώτα πρώτα η διπλή κοινοποίηση. Η κυρία Βαλιά θέλει να αποφύγει όσο είναι και περισσότερο το να αυξηθεί το, το γραφειοκρατικό βάρος. Και επίσης σε σχέση με το πώς απαιτείται να γίνει η κοινοποίηση, εάν αυτές οι επενδύσεις ε, επιβάλλονται από κάποιο συγκεκριμένο νομοθέτημα, τότε τα κράτη-μέλη δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν τα δεδομένα. Αυτό ήδη προβλεπόταν στην πρωτοσκονισμό να χρειαζόταν να ξεκαθαριστεί περαιτέρω. Επίσης κυρία Βαλιάν στέκεται στο, στα θέματα της εμπιστευτικότητας και επίσης ε, της ασφάλειας των δεδομένων σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση και είπε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή να καλύψει και τον άνθρακα για το ενεργειακό μείγμα οπότε και έτσι αυτό να έχει επιπτώσει στην ενεργειακή πολιτική. Άλλο θέμα είναι το κατά πόσο θα πρέπει να καλύπτονται οι επενδύσει ενεργειακή υποδομή σε κάποιε ε, χώρε ε, σε ένα περισσότερο κάτι μέλη και επιπτώσει επίση και ο σύνολο τη Επιτροπή. Και δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι σαν νησί ε, η ενεργειακή μας πολιτική γιατί θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη ότι ισχύει στις γειτονικές χώρες. Επίσης η κυρία Βαλιάν θεωρεί ότι είναι σημαντικό να έχουμε κοινοποίηση των επενδύσεων όσον αφορά κάποια προγράμματα για το φυσικό αέριο, εισαγωγές, εξαγωγές ε, και το ε, υγρό αέριο. Και επίσης είπε ότι που έχουμε με την κατάσταση μικρών σταθμών παραγωγής ενεργειών θα πρέπει να κατέβει το κατόφλι του ορίου της κοινοποίηση. Επίσης είπε ότι θα πρέπει να καλυφθούν και κάποιε εγκαταστάσεις ε, αποθήκευσης λειτουργικής ενέργειας. Περιμένει κύριε Βαλέαν πώς και πώς τη συμβολή συναδέλφων των εισηγητών. Επίσης θα πρέπει ταχύως να διεκπαιρεωθεί αυτό το νομοθέτημα και έχουμε 11 εβδόμου την, ε, την προθεσμία τροπολογίας και το Σεπτέμβριο θα γίνει η ψήφιση στην Επιτροπή. Η ε, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Λάγκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Βαλεάν είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικό ίσως να πετύχει κάποιες προσθήκες και υπάρχει και ένα άλλο σημείο το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Εν γέννη όμως μπορούμε να συμφωνήσουμε στην έκθεση αυτή. Η κυρία Χολ μόλις επεσήμανε ότι υπήρχε διαφωνία προς τη νομική βάση λόγω της ε, πρώην συνθήκης Ευρατόμ θα αποφάσιζε μόνο το Συμβούλιο. Και έκτοτε βέβαια το Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει νέα δικαιώματα έτσι λοιπόν έχουμε και το θέμα της ενέργειας, των μονάδων παραγωγής ενέργειας και της ε, ε, υποχρέωσης κοινοποίηση. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί μιλάμε για τη διαδικασία συναπόφασης και μας δίνει την ευκαιρία να ε, ξαναδούμε τον ε, κανονισμό του 2010 που στηριζόταν στις διατάξεις της Ευρατόμ. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις αυτής της συνθήκης και τις δεσμεύσεις, γιατί ξέρουμε ότι η ενεργειακή πολιτική έχει γίνει ε, κυρίαρχο θέμα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Άρα δηλαδή θα πρέπει να μπούμε και στο περιεχόμενο αυτού του κανονισμού. Έχω να αναφέρω ορισμένα σημεία. Η κυρία Βαλιάνα αναφέρεται και πρότεινε τη συμπερίληψη του άνθρακα. Αυτό το βρίσκω σωστό. Αναφέρομαι στην τροπολογία υπαριθμών 20, την ε, εξόριξη και επεξεργασία του άνθρακα με αιτήσια πραγωγή τουλάχιστον 1 εκατομμύριο τόνους. Ακόμα και εάν ε, θέλουμε να μην έχουμε πια διοξίδι του άνθρακα. Δυστυχώς τον άνθρακα το χρειαζόμαστε ε, για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα. Γι' αυτό και πρέπει να συμπεριληφθεί στον κανονισμό. Μετά, ε, στις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, το αρχικό σχέδιο αναφερόταν ότι θα έπρεπε να γίνεται λόγος μόνο για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Εγώ λοιπόν την εποχή της ε, αποκέντρωσης ε, φοδιασμού με ενέργεια σε ορισμένα κράτη-μέλη, το μέγεθος των εγκαταστάσεων το βρίσκω ή ανεπαρκές ή πολύ ψηλό. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω σε όλα αυτά τα μέτρα να προβλέπετε η μείωση του ε, μεγέθους αναφοράς ανάλογα με την πρόταση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Ε, Παραδείγματος χάρη... Ε, 50 ΜΒ αντί για 100, να λέμε 10 αντί για 20 στη βιομάζα, ε, να μειώσουμε δηλαδή κατά το ίμιση ε, τα μεγέθη, διότι όπως σας είπα θα πρέπει να ανταποκριθούμε στην ε, εποχή της αποκέντρωσης. Επίσης, έχω να αναφέρω και ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά στο άρθρο υπαριθμών 11 Εκεί προτείνεται μία ρήτρα αναθεώρησης ε, στο άρθρο υπαριθμών 11. Αναφέρεται ότι το 2016, το 2016 λοιπόν, η εφαρμογή αυτού του κανονισμού θα επανεξεταστεί, ε, θα κατατεθεί στο ε, Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σχετική έκθεση και μετά υπάρχει μια δεύτερη πρόταση που τη βρίσκω σημαντική, όπου αναφέρεται ότι κατά την επανεξέταση η Κομισιόν εξετάζει την επέκταση εφαρμογής στην ε, εξόριξη ε, εξόριξη ε, και αναζήτηση αερίου, πετρελαίου και εδώ θα περιλάμβανα και το σχιστόλιτο. Πρόκειται για την τροπολογία υπαριθμών 40 ε, για προγράμματα επένδυσης ε, σε τρίτες χώρες. Θα αντέστρεφα λοιπόν την πρόταση της κυρίας Βάλεαν γιατί ε, το κατά πόσον όλα αυτά θα υλοποιηθούν αυτό θα αποφασιστεί, θα κριθεί κάποια στιγμή και ε, ο εφοδιασμός με ενέργεια στην Ευρώπη και αυτό θα κριθεί από το αν θα υπάρξουν αυτοί οι αγωγοί στο νότο της Ευρώπης ή αν θα επεκτείνει το δίκτυό της ε, η Ρωσία. Νομίζω όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν ακριβώς όπως και οι ενεργειακές πολιτικές εξελίξεις σε άλλα μέρη του κόσμου που αναμφίβολα επηρεάζουν ε, τις τιμές. Σας είπα, θα αντέστρεφα την πρόταση της κυρίας Βάλε, αλλά κατά τα άλλα συμφωνώ με όσα αναφέρει στην έκθεσή της. Πολύ ωραία. Ο ε, συνάδελφος κ. Γκλάντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, πολύ σωστά αναφέρατε, σήμερα από ό,τι φαίνεται όλοι εκπροσωπούν όλους. Εγώ μιλάω για τον κύριο Κάμπος ε, που δυστυχώ δεν είναι εδώ. Στην αρχική εισήγηση Αναφέρθηκαν πάρα πολλά και δεν θέλω λοιπόν να επεκταθώ για να κερδίσουμε χρόνο. Η δική μας η πολιτική ομάδα ε, στηρίζει αυτήν την ε, έκθεση. Έχουμε λοιπόν το ενεργειακό ε, σύστημα και καλούμε θα αναλάβουμε μέτρα ενέργειας. Ε, σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με την εισηγήτρια και στηρίζουμε αυτή την ιδέα ε, της ε, κοινοποίησης. Επίσης συμφωνούμε και με την επέκταση των ε, αγωγών σε τρίτες χώρες. Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος κ. Χων, σχετικά με την ε, ε, επικάλυψη των υποχρεώσεων ενημέρωσης, εμείς επιθυμούμε να μην υπάρχει η επικάλυψη αυτή. Επίσης πιστεύουμε ότι η εμπιστευτικότητα των δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν, επειδή τα δεδομένα μπορούν να δημοσιοποιούνται μόνο σε με μια συγκεκριμένη μορφή. Κατά τα άλλα, ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, κάτι το οποίο μέχρι τώρα έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις ε, ε, και οι καθυστερήσεις αυτές παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της αγοράς ε, ενέργειας. Και βέβαια σε άλλες προτάσεις μας θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά όσον αφορά τον σκιώδη συγητή. Προς τον συνάδελφο κύριο Λάγκε να το πω και αν θέλει να με προσέξει. Ε, κοιτάξτε, οι εναλλακτικέ μορφές ενέργειας είναι ένα θέμα που ε, πραγματικά αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Συνάδελφος ε, Τοζανόφσκι. Já teď budu hovořit <laughs> jako stínový zpravodaj, čili θα μιλήσω ως σκιώδης εισηγητής, όχι ως αντικαταστάτης αυτή τη φορά. Επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο συνάδελφος. Νομίζω ότι οι συζητήσεις που έχουμε κάνει στον τομέα αυτό πάνε πραγματικά σε βάθος. Έχουμε εντοπίσει τα, κάποια εφιστάμενα προβλήματα. Από τη μία πλευρά Έχουμε συνέστηση της ε, σημασίας, ε, των στρατηγικής σημασίας δεδομένων στον τομέα της ενέργειας. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι έχουμε ανάγκη πληροφορίες για την ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων. Γιατί το πρόβλημα της Ευρώπης στην ουσία είναι οι συνέργειες μεταξύ των πόρων και το πρόβλημα της διαμετακόμισης. Όσον αφορά τα προβλήματα αυτά, Βεβαίως υπάρχουν και νομικές επιπτώσεις. Στο μέλλον θα πρέπει να αποφεύγουμε τα νομικά προβλήματα στην ε, μετάδοση και ε, διάδοση αυτών των ε, πληροφοριών. Βεβαίως και πρέπει αυτό να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των προϊόντων που θα μελετηθούν. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό του TST τρίτη χώρα, εδώ υπάρχει μια δυσκολία γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα πιο κοντινά γεωγραφικά ε, κράτη που έχουν την ε, μικρότερη απόσταση από την Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρίτες χώρες που επηρεάζουν και θα επηρεάσουν στο μέλλον την ε, ενεργειακή κατάσταση της Ευρώπης, όπως ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες με την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου ή μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές ε, με αυτόν τον τρόπο. Είμαι πεπισμένος ότι η συζήτηση αυτή είναι πιο σύνθετη από ότι η έκθεση που την περιγράφει. Βεβαίως όμως συμφωνώ με την έκθεση και είμαι διατεθειμένος να προσφέρω κάθε βοήθεια ώστε να καταφέρουμε να καθορίσουμε ένα συντονισμό των ενεργειακών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που είναι σημαντικό για τη συνολική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο κύριος Πρόντι τώρα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Κοιτάξτε, ε, κατά την άποψή μου τα θέματα είναι αρκετά πιο σημαντικά, πολύ πιο σημαντικά από ό,τι φαίνεται. Καταρχήν διότι πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση των αναγκών μας σε υποδομές, δηλαδή τόσο των υποδομών μεταφορών όσο και των υποδομών παραγωγής. Άρα με αυτή την έννοια πρέπει να ε, σκοπεύουμε να στοχεύουμε σε ένα σύστημα το οποίο να είναι ε, πραγματικά αποτελεσματικό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι εφόσον μιλάμε για μεταφορές, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η σωστή διάσταση μεταφορών είναι η ευρωπαϊκή διάσταση. Δηλαδή, με αυτή την έννοια θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε, ένα, σε μια αποτελεσματική χρήση, διότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τις πηγές, κυρίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να υπάρχει και μια καλύτερη στατιστική κάλυψη ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε επίσης ε, να έχουμε και καλύτερη χρήση της συντρολεκτρική ενέργειας και μάλιστα με διαφορετικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο από τη αιωλική ενέργεια. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορούμε αφενός να έχουμε αιωλική ενέργεια η οποία είναι προβλέψιμη και από την άλλη έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την υδροελεκτρική ενέργεια όταν δεν υπάρχει επαρκής αιωλική ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οφείλουμε να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις ε, όλης, όλου αυτού του θέματος και οφείλουμε να είμαστε και αρκετά γρήγοροι στο να ε, κάνουμε τις σωστές ε, επενδύσεις. Εδώ λοιπόν για μένα τίθεται και πάλι το θέμα των ευρωομολόγων. Υπάρχουν λοιπόν πηγές, μπορούμε να τις εντοπίσουμε τις πηγές αυτές και με αυτές τις πηγές μπορούμε να έχουμε και αποτελεσματικές μεταφορές. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι με την υψηλή τάση μπορούμε ε, να μειώσουμε την κατανάλωση τρεις φορές σε σχέση με άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Άρα δηλαδή ε, θα πρέπει να μπορούμε να δώσουμε αυτή τη διάσταση στην ηλεκτρική ενέργεια και οφείλουμε να κατανοήσουμε τις αλλαγές που έχουν λάβει η χώρα. Κάτι άλλο θα μπορούσε να είναι και να πούμε και επίσης ε, και για το αέριο, για το δίκτυο αερίου. Ε, δηλαδή και εκεί μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες αποθήκευσης, όπως επίσης και τη δυνατότητα το δίκτυο του αερίου να τοποθετείτε και το αέριο ε, το οποίο παράγεται από τη βιομάζα. Όλες αυτές λοιπόν είναι δικές μου σκέψεις ε, τις οποίες ε, νομίζω ότι μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε γιατί πρόκειται για επίγουσες επενδύσεις οι οποίες μεταξύ άλλων έχουν και τη δυνατότητα να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την ε, οικονομική κρίση. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει απόλυτη προτεραιότητα και θα έχει για τα επόμενα χρόνια. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι η αποθήκευση της ενέργειας ε, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό θεωρώ ότι ε, τα εργοστάσια ε, υδρολεπτικής ενέργειας ε, κατά κάποιον τρόπο είναι ξεπερασμένα. Ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχολεί είναι το εξής. Οφείλουμε να δούμε τον κύκλο ζωής. Δηλαδή τι ακριβώς ε, στοιχίζει ένα ολόκληρο πρόγραμμα από την στιγμή της εγκρισής του μέχρι και την τελική φάση. Και ίσως η Κομισιόν ε, μπορεί να σκεφτεί το θέμα αυτό και θα πρέπει να απαιτήσουμε και εμείς ε, τα βήματα αυτά να γίνονται με απόλυτη σαφήνεια. Και να είναι και επίσης σαφές το που ακριβώς μπορούν να υπάρξουν επενδύσεις, ε, δηλαδή ε, το να υπάρχει ένα πλαίσιο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ε, κεντρικό αίτημα, ένα βασικό θέμα που μας απασχολήσει και στο μέλλον. Άρα δηλαδή στον τομέα αυτό νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και την κυρία Ρόλ που παρουσίασαν πολύ σημαντικά στοιχεία της έκθεσης. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που, για το ενδιαφέρον που δείχνει στο σχέδιο αυτό, για το σχέδιο αυτό κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν θέλει να επενθυμίσει ότι μιλάμε για εφαρμοστικό κανονισμό, ο οποίος ε, παρέχει λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να ενημερώνουν τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επενδύσεις τους. Αυτός ο εφαρμοστικός κανονισμός επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις ανησυχίες που θέτει και η έκθεση. Συγκεκριμένα είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο άνθρακας ήδη συμπεριλαμβάνεται. Έχει περιληφθεί στο παράρτημα της πρότασης κανονισμού αλλά και στον εφαρμοστικό κανονισμό η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνθρακα και οι επενδύσεις που γίνονται στα κράτη-μέλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνθρακα καλύπτονται από αυτόν τον εφαρμοστικό κανονισμό. Αντίθετα, η εξόριξη άνθρακα όπως και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου δεν καλύπτονται και γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει στη ρήτρα αναθεώρησης την δυνατότητα να συμπεριληφθούν και αυτά η γενική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το παρόν είναι ότι προς το παρόν έχουμε μικρή απόσταση από την υλοποίηση του κανονισμού πριν από την ακύρωσή του γιατί μόνο μία έκθεση είχε δημοσιευθεί στις 15 Νοεμβρίου του 2012 τη στιγμή ε, που είχε δοθεί και το σύνολο του πακέτου εσωτερικής αγοράς. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κοινοποιούν κάθε διετία. Όπως ξέρετε ε, ότι ο 617 του 2010 κυρώθηκε αλλά οι επιπτώσεις του εξακολουθούν να ισχύουν, αυτό που καλύπτει εξακολουθεί να ισχύει μέχρι ότου εγκριθεί ο επόμενος. Άρα τα κράτη-μέλη θεωρείται ότι πρέπει να κοινοποιήσουν και πάλι τι επενδύσεις τους φέτος το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το 2014 έκθεση και εμείς σκοπεύουμε να κινηθούμε προς μια ουσιαστική αναθεώρηση του κανονισμού και τη στιγμή που, προβλέπει, που προβλέπεται για την αναθεώρηση να υποβάλουμε μέχρι το Δεκέμβριο 2016 μια έκθεση για την αναθεώρηση, οπότε θα έχουμε ολοκληρώσει τρεις πλήρες περιόδους, ώστε να έχουμε κάποια απόσταση και να ε, ξέρουμε τι πρέπει να τροποποιηθεί και αν χρειάζεται να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή. Αυτό το θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το 2010 στη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο ήδη είχε γίνει πολύ δύσκολο να γίνει πολύ δύσκολα δεκτό ε, να τροποποιηθούν τα κατώτατα όρια των επενδύσεων για τις ανανεώσιμες, Φερρυπίν. Η Κομισιόν προς το παρόν δεν σκοπεύει να ξαναρχίσει αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πρόταση, της οποίας το περιεχόμενο είναι πολύ ε, παρόμοιο με τον κανονισμό του 2010 που ακύρωσε το δικαστήριο και με βάση αυτά που είπε το Συμβούλιο, ε, το Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σε νέα νομική βάση. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θέλω να σας δώσω. Υπάρχουν κάποια πράγματα που σήμερα μας ανησυχούν, όπως Φερρυπίν. Να αποφύγουμε το διοικητικό άχθος στα κρατημέλη, ε, επανάληψη διαφόρων υποχρεώσεων, για τον άνθρακα μίλησα, για τις επενδύσεις με τρίτες χώρες. Ήδη όλα αυτά καλύπτονται από την πρόταση κανονισμού και από τον εφαρμοστικό κανονισμό. Άρα ε, ήδη μπορούμε να το επισημάνουμε. Εν πάση περιπτώσει καλύπτονται αυτά. Όσον αφορά τη διεύρυνση σε νέους τομείς, καλό θα είναι να περιμένουμε τις τρεις εκθέσεις ε, εφαρμογής και να περιμένουμε το Δεκέμβριο του 2006, οπότε προβλέπεται και η αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνει λοιπόν εδώ η συζήτηση και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 12 Ιουλίου το μεσημέρι και κατόπιν στις 2 ε, Σεπτεμβρίου θα έχουμε τη συζήτηση στην Επιτροπή. Ε, πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Μπέλα Κόβας στον σε με συγχωρείτε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επιτροπή, ευχαριστώ όλους για την τροπολογία αλλά και τις προτάσεις σα. Τα βασικά σημεία είναι τα εξή. Έχουμε τώρα την πρόταση αυτή για κοινοτικό σύστημα καταχώρησης των μεταφορών ραδινεργών υλικών. Απευθυνθήκαμε και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, δύναμη του άρθρου 37 του κονζού για να γνωμοδοτήσει όσον αφορά το βάσιμο της αλλαγής της νομικής βάσης αυτής της πρότασης για αυτόν τον κανονισμό για να αντικαταστήσουμε τα άρθρα 31 και 32 ε, ε, που είναι η νομική βάση ε, και επίσης ε, το κεφάλαιο 3 της συνθήκης για της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ατομικής Ενέργειας και είπαμε να προσθεθεί μία διάταξη στη νομική βάση όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η δύναμη του άρθρου 31 αλλά και του άρθρου 32 της συνθήκης Γιουράτων το Κοινοβούλιο είναι το κυρίω αρμόδιο, ενώ δυνάμει του άρθρου 91 το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης με το Συμβούλιο όσον αφορά την συνήθεια νομοθετική διαδικασία. Το συμπέρασμα της Νομικής Επιτροπής είναι ότι το άρθρο 91 αποτελεί την πιο δόκιμη νομική βάση. Είναι το ίδιο συμπέρασμα και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Να αλλάξει δηλαδή η νομική βάση. Τι να δούμε τώρα ως τέτοια το 91. Και επομένως είπαμε και κάποιε προτάσει που λένε ότι θα πρέπει το άρθρο να αποτελεί προσθήκη στην παλιά νομική βάση. Και επίση είπαμε ότι θα πρέπει τώρα να αλλάξει και ο ορισμός για τα κοινά κριτήρια και υπάρχουν και κάποιε άλλε τροπολογίε στον αφορά τον ορισμό του TST, δεν την εγώ υλικό. Επίση, έχουμε κάποιες τροπολογίε για να απαλληφθεί το άρθρο 3, παράγραφο 3, εκεί που λέει ότι Ε, ε, θα πρέπει να δούμε θα γίνει με την ε, οδηγία 96-29 ευρωτών τα βασικά πρότυπα ασφαλεία για αυτού του είδου τα υλικά ή έλεγχο κλειστών πηγών ενέργεια και εκθέτων πηγών σε σχέση με Ιουνίου ακτινοβολίες και θα πρέπει αυτά όλα να καταχωρίζονται ε, όποτε υπάρχει μεταφορά αυτών των ουσιών. Και έχουμε επίσης και ε, κάποιες άλλες που λένε ότι κάθε κράτο μέλος θα πρέπει να ε, διατηρεί το δικαίωμα της απαγόρευση της μεταφοράς ε, ραδιενεργού υλικού στην επικράτειά του εκτός αν ε, έχουμε κάποιο, εφαρμογή κάποιου είδου ε, εθνικές ε, διαδικασίες μεταφοράς και συμφωνώ ότι ο κάθε κάθος μέλος θα πρέπει να αποφασίζει για τον ηλιακό μείγμα του. Οπότε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν τα κράτη-μέλη να ασκήσουν το δικαίωμά τους, να μπορούν να θεσπίσουν αυστηρούς κανόνες σε σχέση με εκείνους που θεσπίζονται με τον ελόγο οργανισμό. Επίσης, συμφωνώ ότι η ο ΔΟΕ μπορεί να προτείνει κάποιους ορισμούς σε σχέση με το πώς θα γίνει η μεταφορά και ποιοι είναι οι καταχωρημένοι μεταφορές. Επίσης, συμφωνώ με την τροπολογία Μαρινέσκου. Ο Μαρινέσκου λέει ότι θα πρέπει να έχουμε μια μεταβατική περίοδο ε, ενός έτους μόλις αρχίσει να ισχύει αυτός ο κανονισμός και έτσι να μπορούμε να έχουμε κάποιο πιστοποίηση όλων των μεταφορέων. Και έχουμε τώρα και κάποιες άλλες τροπολογίες όσον αφορά την περίοδο ε, όπου αυτές οι πιστοποίησεις θα είναι έγκυρες. Κάτι γνώμη μου, μπορούμε να βρούμε μια καλό συμβιβασμό, γιατί δεν απέχουν τόσο, δεν αφήσατε τέλο πάντων αυτέ οι τροπολογίε. Αυτά προ το παρόν. Πολύ ωραία. Το λόγο ε, στο συνάδελφο, στη συνάδελφο Τζόρνταν που αντικαθιστά τον κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ο συνάδελφος μου ζήτησε να παρουσιάσω κάποια από τα βασικά θέματα που ήθελε να θέσει σε σχέση με αυτό τον κανονισμό. Όσον αφορά την νομική βάση, ο κύριος Μαρινέσκου θεωρεί ότι πρέπει να είναι η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πιστεύει ότι πρέπει να καθορίσουμε κοινά κριτήρια για το σύστημα αυτό. Τα κριτήρια πρέπει να στηρίζονται στην οδηγία για την προστασία από την ακτινοβολία και για την μεταφορά επικίνδυνων ουσιών. Κατόπιν ο μεταφορέας μπορεί να πάρει πιστοποιητικό μόνον εφόσον τηρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Τέλος δε, αυτό το οποίο θεωρεί πολύ σημαντικό είναι η πρόσβαση ε, πρέπει να υπάρχει δημόσια πρόσβαση στον κατάλογο των μεταφορέων. Μπορώ να πω και τις δικές μου απόψεις, γιατί αυτά που είπα τώρα είναι αυτά τα οποία είναι η άποψη του κ. Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητήσαμε εκτεταμένα ε, για την νομική βάση του εγγράφου αυτού. Η νομική βάση η οποία επιλέχθηκε, υπερψηφίστηκε, ε, είναι αυτή που προτιμά ο εισηγητής. Η δική μου άποψη είναι λίγο πιο σύνθετη. Διάβασα την γνωμοδότηση Επιτροπής Γιούρη και θεωρώ ότι εκεί έλαβαν υπόψη μόνον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι τις ε, συζητήσεις που είχαμε εμείς στις δικές μας κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εμείς συζητήσαμε για τη θέσπιση κριτηρίων που θα επιτρέπουν την πιστοποίηση ενός μεταφορέα. Τα κριτήρια αυτά είναι πολύ σημαντικά εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, την υγεία των πολιτών από την ακτινοβολία. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ αφενός βοήθειας και προστασίας και αφετέρου ε, διευκόλυνσης της μεταφοράς. Ή ένα από αυτά τα δύο θέματα είναι πιο σημαντικό από το άλλο ή η σημασία τους είναι ίση. Εγώ πιστεύω ότι τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να στηρίζονται στη συνθήκη Ευρατόμ, η οποία στην περίπτωση αυτή τα είναι εξίσου σημαντική με τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλή λοιπόν νομική βάση είναι η καλύτερη επιλογή, η πιο πλήρης επιλογή. Ε, βεβαίως εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά τα έγγραφα, όλα αυτά τα κείμενα θα πρέπει να ψηφιστούν με τη διαδικασία της συναπόφασης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είχαμε και άλλες γνωμοδοτήσεις σχετικές με την κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής, από, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορούν την κοινοποίηση στα κράτη-μέλη. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σωστό τρόπο να μετράμε την αρμοδιότητα του ε, ρυθμιστικού φορέα. Δηλαδή να μην υπάρχει δυνατότητα κάτι να μην πάει καλά εκεί. Με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε ότι από τη Φουκουσίμα κάτι μάθαμε. Ευχαριστώ κυρία Όλπρακ. Like to... Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την τόσο αξιόλογη έκθεση και συμφωνώ ότι θα πρέπει ε, όλοι οι ορισμοί να είναι σαφείς και να συνάδουν προς τα διεθνή ε, πρότυπα και οπότε θα πρέπει πριν ε, ισχύσει αυτή η νομοθεσία να έχουν οριμάσει τα πράγματα τέλος πάντων. Και άκουσα την κυρία Γιορτάνη για την νομική βάση, οπότε θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ θελευρό το, Κοινοβούλιο. Ουσιαστικά δεν έχει λόγο περί αυτού, ε, λόγο των όσων από την Συνδίκη Ευρατών. Έχουμε εδώ τα θέματα υγείας, τα θέματα μεταφορών, περιβάλλοντος. Ε, άρα θα έπρεπε ε, να, εδώ να ισχύει το άρθρο 91 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οπότε εδώ αναδεικνύεται το εξή ζήτημα, ότι η Συνθήκη Ευρατόμ είναι κάτι το ξεπερασμένο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως νομική ε, βάση και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν έχει να κάνει με δημοκρατική νομιμότητα, δημοκρατική λήψη αποφάσεων, διαφάνεια κλπ. Τόσο αφορά την εναρμόνιση των εθνικών ρυθμίσεων ναι, θα πρέπει να υπάρξει συναρμόνιση και έτσι να έχουμε δίκαιες συνθήκες, γιατί αυτό αφορά επίσης την ε, ε, σωστή κατανομή ε, μεταξύ των διαφόρων κατομελών αλλά τελικά μην πάμε για τον ελάχιστο κοινό προγραμμαστή να πάμε για την καλύτερη πρακτική που ισχύει, όπως επιβάλλεται ο πλευράς ασφάλειας. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάθε φορά που θεσπίζεται ένα ε, σύστημα για την Ένωση θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι σε περίπτωση ατυχήματος υπάρχει οικονομική επάρκεια μια που οι συνθήκες θα ήταν πάρα πολύ σοβαρές και επίσης είδαμε τι μπορεί να συμβεί και με το πετρέλαιο όταν μεταφέρεται ε, πόσο σαρωτικέ είναι οι συνέπειε ενό ατυχήματος σε αυτήν την περίπτωση. Οπότε φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει αν έχουμε ατύχημα σε μεταφορά ραδιενεργών υλικών μπορούν να υποστούν τι συνέπειες πάνω από ένα κράτο μέλος. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπε ότι, ότι είναι θέμα κρατών μελών, ε, τα οποία άμα θέλουν μπορούν να καταργήσουν τους ποινικού σταθμού που ακόμα και να απαγορεύσουν τη μεταφορά. Οπότε θα με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας πει αν τα βλέπει όλα αυτά εφικτά. Όσον αφορά τη συμμόρφωση, τι γίνεται όταν κάποιο ε, μεταφορέ, δεν συμμορφώνεται τότε, θα πρέπει και το Επιτροπή να μπορεί να αναστείλει τι δραστηριότητε για λόγου ασφάλεια. Τώρα, θα πρέπει να υπάρχει μια συνοπτική διαδικασία, είναι κάτι γραφειοκρατικό και μακροχρόνιο. Επίση, διαφάνεια στην ελληνική πολύ σημαντική. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωση. κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι όλοι να μπορούν προσβασιμότητα σε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, είναι σημαντικό ε, να γίνεται σε τακτά διαστήματα η αναθεώρηση του οργανισμού μια που θεσπίζει ένα τελείως καινούριο σύστημα την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά στην πορεία θα μάθουμε και θα δούμε αν λειτουργεί εύρυθμα. Ε, καλά όλα αυτά ισχύουν σε κάθε φορά που κανείς θεσπίζει κάτι νέο. Κανείς θα πρέπει να δεχθεί δεν μπορεί να είναι καμία ρύθμιση τέλεια και να επανέρχεται. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι με τη συνθήκη Γιουρετόμη προβλέπεται και το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, και Βεβαίως ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ε, και υπάρχουν διασυνοριακές δραστηριότητες. Το θέμα είναι ε, τι μπορούμε να κάνουμε με τα ραδιενεργά. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και πώς μπορούμε να μεριμνήσουμε Το θέμα είναι επίσης ε, κατά πόσον όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο ζωής. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στον ενεργειακό τομέα να απαλλάξει κανείς ε, τον ενεργειακό, τον τροφοδότη. Συνάδελφο, κυρία Ριβάζη, δεν σας είχα δει που ήρθατε. Έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν για το θέμα αυτό. Εγώ θα επανέλθω στο θέμα της νομικής βάσης. Όπως γνωρίζετε, εδώ και λίγο καιρό στο Αμβούργο, το λιμάνι του Αμβούργου υπήρχε ε, μια πυρκαγιά γιατί υπήρχαν έφλεκτες ουσίες. Έτσι λοιπόν, πώς θα χρησιμοποιήσουμε από τη μία πλευρά μία οδηγία για επικίνδυνες ουσίες ενώ από την άλλη θα χρησιμοποιήσουμε μια οδηγία της Ευρατόμ για τις ραδιενεργές ουσίες. Τώρα όσον αφορά τις, για τις ε, ραδιενεργές ουσίες πετύχαμε αλλαγή της νομικής βάσης. Γιατί λοιπόν για την μεταφορά των ραδιενεργών ουσιών να μην ζητήσουμε ε, αλλαγή νομικής βάσης και να έχουμε δικαίωμα συναπόφασης. Χρειάζεται κάποια συνέπεια σε όλα αυτά. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που θεωρώ πολύ σημαντικό. Πρώτον, η ενημέρωση και η διαφάνεια. Θα πρέπει και οι κοινοί γνώμοι, όπως και οι εργαζόμενοι, να γνωρίζουν τη φύση των ραδιενεργών απορριμμάτων τα οποία μεταφέρονται. Το λέω γιατί γνωρίζω το θέμα προσωπικά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, στους σταθμούς υπήρχαν ραδιενεργά υλικά και το αγνοούσαν, αυτό οι συνδρομικοί υπάλληλοι και πλησίαζαν αυτό και επειδή, επειδή λόγω της ακτινοβολίας έλειωνε το χιόνι πήγαιναν ε, κοντά και στους σταθμούς της NSF πήγαιναν δίπλα σε, αυτούς τους, σε αυτά τα, ε, τα βαγόνια για να προστατευθούν. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο αυτοί που ασχολούνται με την πυρηνική ενέργεια που πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά. Υπάρχουν μια σειρά από άλλους ανθρώπους που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τα υλικά και πρέπει να ενημερώνονται. Όσον αφορά την ασφάλεια, Στην Αλία πρέπει να γνωρίζετε επανειλημμένως μέλη της Greenpeace σταμάτησαν τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών. Είναι άνθρωποι που είναι υπέρ της ειρήνης. Αύριο όμως αν κάποιοι τρομοκράτες σταματήσουν ένα τρένο και χωρί να το σταματήσουν πάνε στο σταθμό μπορούν να πάρουν ραδιενεργές ουσίες. Άρα, όταν υπάρχει μεταφορά σιδηροδρομική θα πρέπει να υπάρξει επαρκής υπηρεσία ασφάλειας και, και να υπάρχει η επαρκή σήμανση και ασφάλεια. Εδώ αυτά τα θέματα δεν τίθεται καν. Κατόπιν υπάρχει και η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Στη Γαλλία όταν γίνεται μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων, ε, ο παραγωγός είναι ο υπεύθυνο, δηλαδή η γαλλική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού, η ΕΝΤΕΦ ας πούμε, είναι υπεύθυνη. Και αν υπάρξει ατύχημα, εγώ θέλω να είναι ξεκάθαρη η ευθύνη. Πρόκειται για τον παραγωγό ή για τον μεταφορέα όταν υπάρξει εκτροχιασμός. Αυτό που έγινε χθες προχθές στον Καναδά. Ποιος έχει την ευθύνη. Ευθύνεται ο μεταφορέας με αυτός που έχει τα βαγόνια ή επειδή υπήρχε το πετρέλαιο εκεί γύρω δεν μπορούσε να υπάρξει επαρκής ε, προστασία. Τώρα, ή ασφάλεις. Θα πρέπει και εδώ να υπάρχει σαφήνεια. Δεν θα πρέπει να τα ψάχνουμε όλα αυτά τη στιγμή του ατυχήματος. Ποιος θα δώσει τις οικονομικές εγγυήσει. Επίσης, οι απάτες. Αν αποκαλυφθεί κάποια στιγμή ότι στη, κατά τη μεταφορά δεν υπάρχουν τα αναφερόμενα ε, ραδιενεργά υλικά, θα πρέπει να απαγορεύεται ο μεταφορέας πλέον να κάνει μεταφορές. Ποιος θα κάνει αυτόν τον έλεγχο. Και αυτό θέτει πρόβλημα. Είναι τα κρατη αυτά τα οποία θα κάνουν τον έλεγχο. Θυμηθείτε ε, τις προειδοποίησεις. Ε, τι θα πει η προειδοποίηση. Θα πρέπει έλεγχος ε, απροειδοποίητος. Και ποιος θα τον κάνει αυτόν τα κρατη Αυτά θεωρώ ότι ε, ο κανονισμός δεν τα καλύπτει επαρκώς. Τέλος, υπάρχει πρόβλημα εναρμόνισης των δοχείων, των κοντέινερ. Υπάρχουν πάσης φύσεως ε, κοντέινερ. Υπάρχουν ε, κάποια που είναι κατασκευασμένα από μπετόν και σε περίπτωση που πέσει αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχουν άλλα, ε, άλλα υλικά που είναι πολύ πιο σκληρά και στα οποία ακόμα και σε σύγκρουση υπάρχει προστασία. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε και το θέμα των κοντέινερ. Έχοντας ελέγξει αυτά τα οποία βλέπουμε, πρέπει να πω ότι ο κανονισμός θα πρέπει να μας προστατεύει και αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Ευχαριστώ η Επιτροπή. Ευχαριστώ ακούνε διάφορα πηγαίνουν για την νομική βάση και ταυτόχρονα να λέτε ότι θα έπρεπε να θεσπιστούν κάποια κριτήρια για αυτού του είδους την αμοιβαία αναγνώριση και την καταχώρηση. Ναι, θα αυτά που να αφορούν τη ραδιοπροστασία, η οποία σαφώς είναι κάτι το οποίο θεσπίζεται, ρυθμίζεται μάλλον μέσω της συνθήκης Ευρατών. Α, ναι, ευχαριστώ λέει και ανοίγει το μικρόφωνο. Ρυθμίζεται λοιπόν από τη συνθήκη Ευρατών και βεβαίως θα γνωρίζετε ότι ε, αυτή είναι lex specialis, επομένως, ειδικό δίκαιο δηλαδή. Και άρα κατησχύει τη γενική ρύθμιση και άρα είναι σωστή η ρυθμική βάση. Και υπάρχει εδώ πέρα μια διάκριση μεταξύ μεταφορέα και μεταφορά. Δεν μιλούμε τώρα για την πράξη τη μεταφορά από το σημείο Α στο Μιλούμε τώρα για τον μεταφορέα. Συγκεκριμένα στο άρθρο 3, παράγραφο 4, ε, λέει με λεπτομέρειε ότι μιλούμε για την πλειοψηφία των μεταφορών και όχι για την εργά πόβλητα ή για κάποιο είδους ε, καύσιμα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ειδική εθνική νομοθεσία. Το σχέδιο δε του οργανισμού αναγνωρίζει ότι αυτού του είδους τα υλικά ε, διέπονται από δική νομοθεσία. Εμείς όμως το λέμε για τους μεταφορείς οι οποίοι θέλουν ή θα ήθελαν να κάνουν τέτοιου μεταφορά. Ας πούμε κάποια φάρμακα, να, δεν χρειάζεται επομένως η αμοιβαία αναγνώριση. Χρειάζεται αυτή η καταχώρηση και μάλιστα να ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Συμφωνούμε επίση 100% με την ε, διαφάνεια. Θα πρέπει να γίνεται, να υπάρχει κάποια δημοσίευση, κατάλογος ε, και εμεί θέλουμε επομένω να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνε για την τιμή συμμόρφωση και επομένω ε, να υπάρχει κάτι σαν blacklist και όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν επίση να προβλέπεται τακτή αναθεώρηση. Εμεί έχουμε ε, συγκροτήσει, έχουμε προτείνει για κάποιο συμβουλευτικό σώμα ε, για την εφαρμογή καθώς και για το λογισμικό που είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μόλις σπιστή νομοθεσία και να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα τροποποίηση. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και επίσης έτσι μπορούμε τώρα να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα. Επαναλαμβάνω ότι εξετάζουμε την περίπτωση των μεταφορέων. Σε περισσότερε περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά για ιατρικέ εφαρμογέ ή για έρευνα και όχι ραδιενεργά υλικά γενικώ. Οπότε, όλα όσα αναφέρονται σε σχέση με την ε, πυρηνική νομοθεσία κάθε χώρα είναι πράγματα άσχετα με την λόγο παρούσα συζήτηση. Πολύ ωραία. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Ε, το λόγο στην... Ε, στον Μπέλα Κόβατς. Σας ευχαριστώ, Αξιότιμη κύριε βουλευτέ. Ε, επίσης ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά τα οποία αναφέρθηκαν στη σημερινή συζήτηση και οπωσδήποτε θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη και εγώ έχω την πεποίθηση ότι όπως και άκουσα από τους συναδέλφους σε κάποιο σημείο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο κοινό παρανομαστή. Το πιστεύω αυτό. Και μόλις καταλήξουμε και μόνο το συντομότερο που θα, τα συμφωνήσουμε τόσο το καλύτερο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να επενθυμίσω στους ε, συναδέλφους ότι θα ψηφίσουμε στις 18 ε, Σεπτεμβρίου. Τελειώσαμε λοιπόν τις εργασίες μας. Η συνεδρία της Επιτροπής θα συνεχιστεί αύριο στις 9 το πρωί και έτσι λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στη συνεδρία των συντονιστών σε λίγα λεπτά. Σε λίγα λεπτά.